Colleagues, uh, please take your seats and we'll get started. για να ξεκινήσουμε. Το πρώτο θέμα στην ε, στην διάταξη προβλέπει να σας πω ότι είμαι εισηγητής αλλά προεδρεύω τη απουσία του Προέδρου Φερνάντο Λόπες Αγγιλάρου αλλά και οι αντιπρόεδροι μας ε, αδυνατούν να παρευρεθούν ως εκ τούτου θα προεδρεύσω εγώ σήμερα το απόγευμα. Θα σας πω καταρχήν, επειδή έχουμε μια μικρότερη αίθουσα σήμερα, έχουμε με διερμηνία μόνο τα γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά, ουγγρικά, πολωνικά και ελληνικά. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν ε, αν κάποιοι δεν έχουν διερμηνία στη γλώσσα τους. Περνάμε στην 8η ακρόασή μας. Δύσκολο να φανταστούμε ότι έχουμε ήδη κάνει 7 ακροάσεις. Αυτή, όπως είπα, είναι η 8η και έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Μέχρι τώρα είχαμε κάποιες καλά οργανωμένες ακροάσεις που εστιάζαν στη νομική δουλειά και αφορούσαν ιδιαίτερα την κατάσταση στις ΗΠΑ. Σήμερα θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στην νομική κατάσταση σε διάφορα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εθνικό επίπεδο, ενωσιακό επίπεδο, επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης και επίπεδο διεθνούς δικαίου. Σήμερα θα δούμε και κάποιες εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις που ενδιαφέρουν όλους όσοι θα ακούσουν σήμερα, είτε παρίστανται εδώ, είτε μέσω το web streaming. Θα σας ε, αναφέρω τους αγορητές, αλλά πριν από τις τρεις παρουσιάσεις θα ήθελα να σας εξηγήσω πως λόγω του ότι πιέζει ο χρόνος και έχουμε προσθέσει και έναν ακόμα μιλτή στο δεύτερο τμήμα των εργασιών μας θα μάλλον μετά τις παρουσιάσεις θα ακούσουμε τους κοιόδης και εμένα ως εισηγητή, καθώς επίσης και ερωτήσεις από κάποιους που θα θελήσουν να θέσουν ερωτήσεις. Συμφωνείτε? Δεδομένου ότι υπάρχει ένας μόνος κοιόδης στην αίθουσα, ε, συμφωνεί πάντως, εντάξει. Άμα συμφωνείτε εσείς. Θα συζητήσω λοιπόν με τον ένα εκ των συντονιστών, εντάξει κύριε Βόσο. Μια του ότι εσείς μόνο είστε παρόν, ούτως θα λειτουργήσουμε. Όπως σας είπα θα εστιάσουμε τώρα σε τρεις παρουσιάσεις που αφορούν διάφορα νομικά ζητήματα και να δούμε κατά πόσο τα θεμελιώδη δικαιώματα έχουν παραβιαστεί σε σχέση με τις δραστηριότητε παρακολούθησης Καταρχήν, ο ε, διεθνής νόμος, ε, το ενωσιακός νόμος ε, και ο ΕΣΔΑ. Πρώτος, ο συνάδελφος θα μιλήσει για διεθνές δίκαιο, είναι καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ήταν ειδικός στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο καθηγητής Σέναν είναι επίσης επικεφαλή του προγράμματος Survey που χρηματοδοτεί το 7ο, πλαίσιο, 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ο πλαισιο προγραμμα Σουάνων θα καλύψει το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Κύριε Σουάνων, έχετε το λόγο και μπορείτε να μιλήσετε επί 10 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ. Σε ερώτημα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παρευρίσκομαι σε αυτήν την αξιότιμη επιτροπή για να συζητήσουμε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα, όπως σας εξήγησε και ο Πρόεδρος. Εγώ θα καλύψω τα ζητήματα διεθνούς δικαίου ως προς το κατά πόσον η ηλεκτρονική παρακολούθηση την οποία διεξήγαγαν οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο κυρίω συνιστούν παραβίαση του διεθνού δικαίου. Πρώτα απ' όλα τίθεται το θέμα τη νομιμότητα. Πολλέ χώρε συμμετέχουν και συνεχίζουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966 που είναι ένα από τα σημαντικότερα ε, νομικά κείμενα των Ηνωμένων Εθνών, που έχει κυρωθεί από 196 χώρες στον κόσμο και ε, εν πολλής είναι και ένα σύμφωνο το οποίο προηγήθηκε και ενέπνευσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ούτω, ούτω ούτε οι Ηνωμένε Πολιτείε ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν δεχθεί τη δυνατότητα υποβολής ατομικών προσφυγών με βάση το σχετικό πρωτόκολλο. Κάτι που θα είχε επιτρέψει στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ να διεξάγει έρευνες και να ε, εξακριβώσει κατά πόσον παραβιάστηκαν τα ατομικά δικαιώματα ενός προσφεύγοντα. Ωστόσο, υπάρχει δυνατότητα ε, παρέμβασης της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε γενικό επίπεδο για να εξετάσει κατά πόσον το σύμφωνο γίνεται ε, σεβαστό και αυτό γίνεται με βάση το άρθρο 41 του συμφώνου. Δεν έχει αναλυφθεί μέχρι τώρα μια τέτοια πρωτοβουλία, μια τέτοια διαδικασία δεν έχει ξεκινήσει. Αυτό που διαπιστώνουμε ότι δύο δυτικές δημοκρατίες έχουν παραβιάσει, έχουν παραβιάσει σε μαζικό επίπεδο τα ατομικά δικαιώματα και την ιδιωτικότητα εκατομμυρίων πολιτών, ευρωπαϊκών πολιτών. Επομένω, αυτή η διαδικασία προσφυγής θα έπρεπε να ή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ταυτόχρονα με βάση το σύμφωνο αυτές οι δύο χώρες είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν περιοδικές εκθέσεις στην Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τις οποίες εξετάζει και, και ε, αποφασίζει κατά πόσον υπήρξε ε, συμμόρφωση ή όχι με το σύμφωνο. Την εβδομάδα αυτή αναμένεται η υποβολή της περιοδικής εκθέσης των ΗΠΑ και του ΗΠΑ του χρόνου. Το επόμενο θέμα είναι κατά πόσον οι δραστηριότητες ηλεκτρονικής παρακολούθησης των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν παραβίαση του άρθρου 47 του ICCPR. Ο λόγος που αποτελούν ε, παραβίαση είναι επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα ατομικής προσφυγής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να ε, εξεταστεί το θέμα στο επίπεδο της Επιτροπής. Λοιπόν, όλα τα κράτη-μέλη έχουν το θετική υποχρέωση να δημιουργήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα προστατεύει την ιδιωτικότητα και το απόρριτο των επικοινωνιών και να προστατεύσουν τους πολίτες από τέτοιες ε, παραβιάσεις ανεξαρτήτως εάν αυτές οι επιθέσεις της ενάντια στην ιδιωτικότητά τους προέρχονται από ιδιώτες είτε από το κράτος. Το 1988 υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ένα γενικό σχόλιο το οποίο ερμηνεύει το σύμφωνο. Συνήθως τέτοιου γενικά σχόλια ε, αντλούν από τις αποφάσεις που ελήφθησαν επί ατομικών προσφυγών ή τις εξετάσεις των περιοδικών εκθέσεων το 88 η εμπειρία που είχε συσσωρευτεί ήταν κάπως περιορισμένη. Επομένως δεν θα μπορούσε κανείς να αναμένει ότι όλα τα ζητήματα του απορρίτου και της ιδιωτικότητας θα μπορούσαν να έχουν ληφθεί υπόψη. Έχω εδώ διαλέξει δύο παραθέματα από αυτό το γενικό σχόλιο. Πρώτα απ' όλα γίνεται σαφές, σαφής μνήα στο γεγονό ότι χρειάζεται νομική βάση προκειμένου να αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών, καθώς επίσης και το γεγονό ότι ήδη από το 1998 καλύπτονταν οι βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι υπολογιστές. Ο ειδικό, ανταποκριτή ε, για την ε, τρομοκρατία από το 2005-2006, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που είναι ξεχωριστό όργανο του ΟΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξέδωσε ένα πόρισμα μια θεματική έκθεση που αφορά το δικαίωμα στο απόρριτο των επικοινωνιών στο πλαίσιο του πολέμου κατά τη τρομοκρατία, η οποία εξετάστηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Μάρτιο του 2010. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, εξέτασε την πιθανότητα να αποσύρει το σχόλιο του ε, για το Γενικό Σχόλιο 16 και να το αντικαταστήσει με ένα καινούργιο Γενικό Σχόλιο που θα λαμβάνει απόψε τις εξελίξεις που συνέβησαν στο μεταξύ. Ως ειδικό ανταποκριτή λοιπόν για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της τροποκρατίας, ε, εγώ βασίστηκα αφενός στο σχόλιο 16 τη γενικότερη πρακτική για τις πολιτικές που είχε υιοθετήσει η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εν τω μεταξύ και το αποτέλεσμα αυτής της ε, εργασίας ήταν η δημιουργία ενό, μιας δοκιμασίας, ενός τεστ, ενός καταλόγου των προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται για να θεωρείται αποδεκτή η άρση του απορρίτου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα συνιστά παραβίαση του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. ο πυρήνας κάθε ανθρώπινο δικαιώματος, όπως το απόρριτο των επικοινωνιών, είναι απαραβίαστο και σε περίπτωση που, θα, που υφίσταται η δυνατότητα άσκησης της κριτική ευχέρειας στην, ε, ε, εφαρμογή αυτού του δικαιώματος, η, ε, η περιορισμός του δικαιώματος θα πρέπει να γίνεται με, κατά τρόπον αναλογικό. Θα πρέπει να επιλέγεται η λιγότερο παρεμβατική μέθοδος και θα πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστή η αρχή της αναλογικότητας κατά τη στάθμιση των δύο ένωμων αγαθών. Επίσης, η άρση του δικαιώματος στο απόρριτο δεν θα πρέπει να οδηγεί σε άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι σωρευτικές. Πρώτα απ' όλα, η αρχιτεκτονική, το οικοδόμημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, η οποία κατάρτισαν, δημιούργησαν οι Ηνωμένε Πολιτείες, παραβιάζει Ορισμένε από τι ρήτες, ορισμένα από τα στοιχεία αυτής της δοκιμασίας. Και με βάση αυτό θεωρώ ότι έχει υπάρξει ε, παραβίαση του άρθρου 17 του ICPR. Με άλλα λόγια, θεωρώ ότι η ηλεκτρονική παρακολούθηση από τις ε, ε, ΗΠΑ αποτελεί αυθαίρετη παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα. Μια και δεν έχω πολύ χρόνο στην διαθεσή μου, θα αναφερθώ μόνο σε ορισμένα από αυτά τα στοιχεία που την καθιστούν παράνομη την παρακολούθηση. Πρώτον, δεν βασίστηκε σε υφιστάμενη νομοθεσία, όπως θα έπρεπε με βάση το δίκαιο ανθρωπινών δικαιωμάτων, βασίστηκε ανταυτού στην, ε, ε, στην νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία των μυστικών υπηρεσιών και την καταπολέμηση της τοποκρατίας βασίστηκε επίσης σε νομολογία που δεν επιτρέπει στα άτομα να ε, λάβουν τις αποφάσεις τους με βάση δεδομένα δημοσίως διαθέσιμα. Επίσης ο συστηματικός χαρακτήρας της συλλογή των μεταδεδομένων δημιουργεί ανησυχίες, γιατί όσο πιο συστηματική είναι αυτή η ανάλυση, τόσο περισσότερο ενέχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε μια κατηγοριοποίηση η οποία τελικά είναι φωτογραφική. Άρα δεν υπάρχει ε, ε, σεβασμός του δικαιώματο του, της ιδιωτικότητας. Εξάλλου τα μετοδεδομένα απλώ χρησιμοποιήθηκαν ω ενδιάμεσο στάδιο πριν να εξαχθούν και να αναλυθούν προσωπικά δεδομένα ως μέρος του ιδίου του περιεχομένου. Ορισμένα από αυτά τα ζητήματα μας έχουν απασχολήσει στο πλαίσιο του προγράμματος Survey, που αναφέρατε και εσείς κύριε, κύριε Πρόεδρε. Στο φάκελο που σας διανεμήθηκε έχουμε, ε, ε, σας έχουμε δώσει κάποιες φωτοτυπίες από το υπόδειγμα που χρησιμοποιούμε, υπόδειγμα αξιολόγηση. Είναι ένας πίνακας αξιολόγησης των διαφόρων τεχνικών παρακολούθησης βασίζεται σε δύο παράγοντες κυρίως. Τη σημασία ενός θεμελιώδους δικαιώματος σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αφενός και αφετέρου σε ποιο βαθμό ε, υφίσταται παραπεριορισμός σε αυτό το δικαίωμα. Η οποία αναλύεται ως σε δύο ε, στοιχεία, το κατά πόσον υπήρξε νομική ε, εξουσιοδότηση, καθώς επίσης και τη διάρκεια της παρακολούθησης. Προσπαθούμε να αξιολογήσουμε την, τον πρόοδο της τεχνολογίας και να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό οι νέες τεχνολογίες παραβιάζουν τον πυρήνα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς δεοντολογίας, από πλευράς νομικής και καταλήγουμε σε ένα είδος βαθμονόμησης ε, με τρία επίπεδα, το πράσινο, το κίτρινο και το κόκκινο. Στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, πέρα από το, ε, την έκδοση Γενικού Σχολείου με βάση το άρθρο 17 του ICCPR, η Γερμανία ανέλαβε μια πρωτοβουλία να προτείνει ένα νέο πρόσθετο πρωτόκολλο στο ICCPR τη μελετάμε αυτή την πρωτοβουλία, αλλά αυτή δεν υποβαθμίζει τη σημασία της εφαρμογής του υφιστάμενου διεθνούς δικαίου και της αξιολόγησης των δραστηριοτήτων παρακολούθησης με βάση το υφιστάμενο δίκαιο. Συμπερασματικά έχουν σειρά συστάσεων. Πρώτα απ' όλα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκδώσει μια έκθεση. Την επόμενη εβδομάδα αναμένουμε την αξιολόγηση της περιοδικής έκθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ, θα μπορούσε το, Ηνωμένο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο να υποβάλει στον ΟΗΕ ε, προσφυγή κατά των Ηνωμένων Πολιτειών ως προς ε, την παραβίαση του άρθρου 17 του ICCPR. Επίσης θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί η πρωτοβουλία της Γερμανίας για ένα νέο πρόσθετο προαιρετικό πρωτόκολλο στο ICCPR. Καθώς επίσης θα πρέπει να ενταθούν και οι προσπάθειες για την, την εξέταση του συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και ιδιαίτερα της ε, κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών της GCHQ στη συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να κατά την άποψή μου να συνεχίσει να υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών και της ιδιωτικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σένιν, και ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε το χρονοδιάγραμμα. Να επαναλάβω ότι όλη η παρουσίαση έχει ανέβει στην ιστοσελίδα του EpiWeb. Οπότε όποιος θέλει να δει την πλήρη παρουσίαση μπορεί να τη βρει εκεί. Θα αρχίσω τώρα με τους ασκαιώδεις εισηγητές. Αρχίζει ο κύριος Φως. Αγαπητέ κύριε Σένιν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ακούσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για την ε, σύμβαση αυτή. Ε, ορισμένες ερωτήσεις έχω σχετικά με το Σύμβαση Δικαιωμάτων. Ε, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη για τους επικούς τρίτων χωρών, εθνικούς υπήκους προστασία των πολιτών μιας χώρας η οποία διεξάγει ε, τέτοιες ε, δραστηριότητες. Επιπλέον, μια άλλη ερώτηση. Ε, παραβίαση αποτελεί μόνο η αποθήκευση δεδομένων ή και η ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων αυτών. Και αναφέρατε ήδη κάτι γενικότερο για το άρθρο 17. θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι συνέπειες μιας ε, εθνικής προσφυγής. Ποιες συνέπειες υπάρχουν για τους ε, πολίτες και σε γενικότερο ε, πλαίσιο, ότι είναι δυνατόν ποιο όφελος έχουν οι πολίτες και ποιες είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας προσφυγής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βός. Κύριε Άλμπρεχτ έχει το λόγο. Πρώτα θα υποβληθούν όλες οι ερωτήσεις. Και κατά κάποιο μαγικό τρόπο όλοι τηρείτε στο το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό. Αλλά η παρουσίαση ήταν στα χρονικά όρια που προβλέφθηκαν και οι ερωτήσεις επίσης. Κύριε Άλμπρεχτ, ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ σημαντική παρουσίαση. Σαφώς υπάρχουν παραβιάσεις ή δυνατές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και καμία κυβέρνηση δεν το τονίζει αυτό. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το ότι μια κυβέρνηση, κάποιος διεθνής οργανισμός διερευνά αυτήν την στιγμή αυτές τις ε, πιθανές παραβιάσεις. Και όσον αφορά τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών, εσείς τι αναμένετε να γίνει σε πολιτικό επίπεδο. Διότι φυσικά και αυτό είναι κάτι το οποίο τα Εθνικά Κοινοβούλια και εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Και μια τελευταία ερώτηση τώρα από τους ασκιώδους και από εμένα είναι ότι, κύριε καθηγητά Σένιν, αναφέρατε ότι η Επιτροπή των ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνεδρίασε στην Γενέβη για το θέμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεδριάσει. Μπορείτε να μας πείτε ποιο αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα. Θα δεχτούν οι Ηνωμένε Πολιτείε τις συστάσεις των Ηνωμένων Δεθνών σε σχέση με το άρθρο 17 του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Ποιες είναι οι προσδοκίες σας ή μια πολιτική ανάλυση. Μόλις απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις ε, μου υποβλήθηκαν. Καταρχάς, ε, κύριε Φως, το σύμφωνο δεν διαχωρίζει σε πολίτες και μη πολίτες. Είναι πολύ σπάνιο να αναφέρονται τα πολιτικά δικαιώματα μόνο των ε, πολιτών. Δύο είναι τα σχετικά δικαιώματα. Πρώτον, το δικαίωμα συμμετοχής του άρθρου 25, το οποίο αναφέρεται μόνο σε πολίτες σε εθνικό επίπεδο και το δικαίωμα ενός πολίτη να μην απελαθεί από τη χώρα του. Η διασυνοριακή μετακίνηση έχει διαφορετικές προποθέσεις για ε, πολίτες μιας χώρας και για μη πολίτες μια χώρας. Τώρα υπάρχει και το εδαφικό αντίκτυπο του Διεθνούς Συμφώνου οι επιπλοκές και, τα, και επιπτώσεις εκτός ε, συνόρων της Ευρώπης. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από την αρχή έχει απορρίψει αυτές ε, τις ε, θεωρήσεις αρχίζοντας από την περίπτωση Μπούργκος στην Ουρουγουά. Ίσως αυτή είναι η πιο γνωστή περίπτωση. Η Επιτροπή ήταν ξεκάθαρη στη διατύπωση δηλώσεων δεν είχε σημασία πού σημειώθηκε η παραβίαση, σημασία είχε το αποτέλεσμα, η παραβίαση δηλαδή του συμφώνου. Ακόμα και αν ε, αυτή η παραβίαση συμβαίνει εκτός εθνικών συνόρων, συμπεριλαμβάνεται και θεωρείται παραβίαση του Διεθνούς Συμφώνου. Και αυτό είναι σαφές στο σύμφωνο, στο άρθρο 17 τώρα. Μία άλλη ερώτησή σας ήταν οι συνέπειες μιας παραβίασης. Πράγματι, η διαδικασία προσφυγής είναι ένα μέσο που γίνεται αποδεκτό στα Ηνωμένα Έθνη σε περίπτωση που ένα κράτος ε, δεν έχει κάνει δεκτή μία ατομική προσφυγή. Υπάρχουν μηχανισμοί προσφυγής σε 113 ε, χώρες. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία των, ε, της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Οι Ηνωμένε Πολιτείες όμως και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν υπογράψει ε, κάποια τέτοια συμφωνία. Δεν ξέρω βέβαια τι συζητιέται στους διπλωματικούς κύκλους, αλλά υπάρχουν ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής οι οποίες συζητούν το ενδεχόμενο τέτοιας προσβυχής και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Φυσικά υπάρχουν και οι ορισμένες δυνατότητες στα πλαίσια του ε, Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου. όπου κάτι μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση διεθνούς δικαίου και όχι κάποιες εθνικής Σε Τέλος, όπως είπα, στην συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα εξετάσουμε την έκθεση για τις Ηνωμένε Πολιτείες και ο πρόεδρος με ρώτησε τι αναμένω προσωπικά από αυτήν την συνεδρίαση. Θα γίνουν κάποιες συμπερασματικές ε, παρατηρήσεις ε, την 1η Νοεμβρίου από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή έχει υποβάλει ορισμένες ερωτήσεις, την επιτροπη ανθρωπινων δικαιωματων η επιτροπη εχει υποβαλει ορισμενες ερωτησεις την υπαριθμόν 22 αλλά και άλλες σχετικές με την ε, δομή της NSA και της δραστηριότητας παρακολούθησης της. Ίσως αναμένουμε μία δήλωση ασυμβατότητας με το άρθρο 17 αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ποια θα είναι η έκβαση της συνεδρίασης. Τώρα, κύριε Βός, ε, με ρωτήσατε εάν η απλή αποθήκευση δεδομένων καθιστά παραβίαση. Ενδεχομένως, ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ευρύ φάσμα μεθόδων παρακολούθησης, μια αρχιτεκτονική δομή που αποτελείται από πολλά επιμέρους στοιχεία. Και ναι, στο σύνολό τους αυτέ οι δραστηριότητε καθιστούν παραβίαση του άρθρου 17, όμως το σημείο αυτό που βρισκόμαστε τώρα εξετάζουμε την, ε, αποθήκευση, την σκόπιμη αποθήκευση δεδομένων για σκοπούς εξέτασης ε, μεταδεδομένων που σχετίζονται με πολίτες και έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσβαση με τα δεδομένα. Αυτό καθιστά παραβίαση του άρθρου 17. Νομίζω πως απάντησα και στον κύριο Άλμπρεχτ και για το τι κάνουν οι άλλες χώρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Κύριε Φως. Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Έχω κάποιες ε, μικρές ερωτήσεις. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει μια τέτοια συλλογική προσφυγή επιπλέον. Πιστεύω πως και εσείς λαμβάνετε παρόμοιες πληροφορίες όπως εμείς από τον τύπο, όπου δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση για τις δραστηριότητε ε, αυτές. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς διαπιστώνετε ότι όντως έχει ε, υπάρξει παραβίαση του άρθρου 17. Βασίζεστε μόνο σε δηλώσεις τύπου, σε συνομιλίες με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι όντως έχουν αποθηκευτεί δεδομένα ή όχι. πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίζεστε. Ποιο είναι αυτό. Απαντώντας την πρώτη ερώτηση, θα ε, να πω ε, πως ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, είναι μέλος της ICCPR Βρισκόμαστε λοιπόν στα χέρια των ε, μεμονωμένων κρατών. Τώρα το θέμα είναι αν υπάρχουν αρκετέ αποδείξει. Νομίζω πως υπάρχουν. Εφόσον οι ΗΠΑ πολιτείες καλύτερα από το ΙΤΑΒ δέχονται την ύπαρξη κάποιων στοιχείων για τα προγράμματα αυτά παρακολούθησης. Ε, έχουμε κάποια βασικά στοιχεία όπως ε, το έχουν δηλώσει αρμόδιες αμερικανικές αρχές. Γνωρίζουμε τις διατάξεις επίσης του Foreign Surveillance Act και την νομική βάση. Ξέρουμε πόσο ασαφές όργανο είναι και είναι αδύνατον ε, για τον πολίτη να κατανοήσει ποια θα είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Επίσης ε, υπάρχει για μένα μια, ένα μυστικό δικαστήριο και μια ε, μυστική διαδικασία. Επίσης γνωρίζουμε ότι και τα εποπτικά όργανα του Κογκρέσου και το ε, ε, δήλωσαν ότι απέτυχαν στην εποπτεία τους. Το κριτήριο δηλαδή που προβλέπει ο νόμος και οι νομικές απαιτήσεις που χρειάζονται έχουν αποδειχθεί. Υπάρχει πάντως ε, έλλειψη νομικής βάσης. Ευχαριστώ. Παρακαλώ κυρία Σίπουλα για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποβάλει μια προσφυγή. Μπορούμε δηλαδή εμείς ε, να υπογράψουμε το Διεθνές Σύμφωνο και μετά να ε, προσφύγουμε. Θα ήταν και αυτό μια νέα οδός. Έπειτα, οι παραβιάσεις αυτές ε, του άρθρου 17 για την ε, εισφολή στην ιδιωτική ε, ζωή των πολιτών ε, δικαιολογούνται πάντα ως θέμα εθνικής ασφάλειας και αυτοί οι μηχανισμοί παρακολούθησης δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσως δεν είναι απόλυτα δική σας αρμοδιότητα, αλλά έχετε να μας πείτε κάτι σχετικά με την διαδικασία, εάν η διαδικασία αυτή η προσφυγή σε μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ε, διεθνή νομολογία και να επηρεάσει την ε, διεθνή νομολογία σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει κίνδυνος για το κράτος δικαίου έτσι όπως το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Σένσιου έχει μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Στην έκθεσή σας από το 2009 για την προώθηση και προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών υπό το πρίσμα της αντιτρομοκρατίας αναφερθήκατε στο δικαίωμα της ιδιωτικότητας στα πλαίσια της μάχης κατά της τρομοκρατίας σε σχέση με τις ε, Δυνατότητε παρακολούθησης. Αυτά τα μέτρα όχι μόνο απειλούν το δικαίωμα των πολιτών στην ιδιωτικότητα, αλλά και επηρεάσουν την ελευθερία κίνηση, ιδιαίτερα στα σύνορα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Τέσσερα χρόνια μετά, ποιες θεωρείτε ε, ότι είναι οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της αντιτρομοκρατίας οι οποίες απειλούν τα, το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών και επιπλέον πώς αξιολογείτε εσείς την αποτελεσματικότητα της συλλογής δεδομένων για τη μετακίνηση των ε, πολιτών στα πλαίσια της ε, αντιτρομοκρατίας. Και τέλος, ποιες ε, νομικές ασφαλιστικές δικλείδες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απειλής της ενδιωτικότητας στα πλαίσια του, των διασυνοριακών ελέγχων, ιδιαίτερα εν ώψη των αυτοματοποιημένων ε, διασυνοριακών ελέγχων και όσον αφορά την, ε, την ε, διαχείριση των συνόρων. Τι έχει ακόμα εφαρμογή σήμερα από αυτά που έγιναν το 2009. Και μια τελευταία ερώτηση από τον Άξελ Φως. Να με συγχωρείτε που πάντα παίρνω το λόγο σε τμήματα. Να πω βέβαια ότι εσείς μα λέτε ότι το άρθρο 17 αναφέρεται σε ε, ενέργειες παρακολούθησης και διαπιστώνονται παραβιάσεις, ηλεκτρονικές παραβιάσεις ε, παραβιάσεις ε, μέσω της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Ε, πού είναι όμως τα όρια ανά στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα. Πού βρίσκονται τα όρια λοιπόν της ιδιωτικότητας από τη μία και, και του κινδύνου και για την εσωτερική και εθνική ασφάλεια και ενός γενικότερου κινδύνου. Ευχαριστώ πολύ μπορείτε να δώσετε τις τελικές απαντήσεις και τα συμπερισματικά σας σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αρχίζω από τον κύριο Βός. Πράγματι, η αντιτρομοκρατία είναι μία ανάγκη και αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν και αυτές τις εισβολές στην ε, ιδιωτικότητα. Πού λοιπόν ε, υπάρχουν τα όρια, ρωτήσατε. Μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της ε, συλλογής δεδομένων όπου οι πάροχοι μπορούν να αποθηκεύουν δεδομένα από 6 έως 12 μήνες και μόνο μετά από συγκεκριμένη έγκριση, κατόπιν απόφασης, οι αρχές έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Αυτό μπορούμε να το θεωρήσουμε ασφαλή μέθοδο, αλλά ακόμα και αυτή η μέθοδος είναι αμφιλεγόμενη στην Ευρώπη. Διότι υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν τους 24 μήνες υπερβολικά, μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι θεωρούν πως ε, δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις ε, εταιρείε για την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων, ότι πάντα μπορούν να υπάρξουν παραβιάσεις. Πιστεύω όμως πως έχουμε επιλέξει μία μέθοδο η οποία βασίζεται σε διεθνή νομοθεσία. Και μέθοδο σε αυτή μας δίνει μεγαλύτερη δυνατότητα πρόβλεψης από ότι για παράδειγμα η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη, η διαδικασία έγκρισης χρειάζεται αυστηρότερο έλεγχο. Πρέπει να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι προϋποθέσεις ε, κάτω από τις οποίες οι αρχές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Εδώ δίνεται ιδιαίτερα βάση στο, σε ένα σύστημα δικαστικής έγκρισης, διότι ένα τέτοιο σύστημα θα μειώνει τις επιθανότητες παραβίασης ή εισβολής στην ιδιωτικότητα. και ως κατά συνέπεια θα αποτελεί παραβίαση των ε, θεμελιδών δικαιωμάτων. Η κυρία Σίπελ μας ρώτησε αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στο σύμφωνο. Δυστυχώς όχι. Οι συνθήκες αυτές έχουν συνταχθεί έτσι ώστε μόνο κράτη να μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτές. Η μόνη εξαίρεση είναι, η, είναι το σύμφωνο για την αναπηρία, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση για πρώτη φορά είχε τη δυνατότητα να υπογράψει την σύμβαση αυτή. Οτιδήποτε άλλο θα χρειαζόταν διαδικασία τροποποίησης που είναι βέβαια πιθανό ενδεχόμενο, όμως ε, θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να πραγματοποιηθεί. Μετά, όσον αφορά το, τον αντίκτυπο άλλων ε, περιπτώσεων και την απειλή για το κράτος δικαίου, πιστεύω πως είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται μεγάλη προσοχή ιδιαίτερα ε, από τον ε, νομικό κλάδο, από τους, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ε, τους ευρωβουλευτές. Πιστεύω πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εάν γίνει γενικά αποδεκτό το ότι η ιδιωτική ζωή πλέον δεν υφίσταται και δεν υπάρχει ιδιωτικότητα, τότε ενδεχομένως αυτό να έχει ένα, ένα αντίκτυπο και σε άλλα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια περίπτωση και χρειάζεται την δέουσα προσοχή. Όχι μόνο ε, για τη συγκεκριμένη παραβίαση, αλλά και για τις ε, επερχόμενες ενδεχόμενες παραβιάσεις. Τώρα, κύριε Έντσιου, ε, μας ρωτήσατε για τη διασύνδεση των δικαιωμάτων, το δικαίωμα της ε, ελεύθερης μετακίνησης και των διασυνοριακών ελέγχων και το πώς η ελευθερία της κίνησης επηρεάζεται έμεσα από τις νέες τεχνολογίες παρακολούθησης, τις βάσεις δεδομένων κτλ. Και τα λεγόμενα έξυπνα ηλεκτρονικά σύνορα. Αυτό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός ε, τομέας, ο οποίος χρειάζεται προσοχή στα, πλαίσια, γενικότερα πλαίσια της παρακολούθησης μπορούμε να δούμε ότι η παρακολούθηση αυτή πρωτίστως ε, έχει επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα. Υπάρχουν όμως και έμεσες επιπτώσεις σε άλλα ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαίωμα ελεύθερης συνάθρησης, ελευθερίας της έκφρασης, ανεξιθρησκεία. Όλα αυτά επηρεάζονται εμέσως. Μετά μπορούμε να μιλήσουμε για ένα μια έμεση επίπτωση, το chilling effect, όπου οι πολίτες δεν τολμούν μετά να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα, γιατί φοβούνται ότι οι κινήσεις τους παρακολουθούνται. Και αυτό έχει επιπτώσει σε πάρα πολλούς τομείς, σε, σε ποιες ε, θρησκευτικές οργανώσεις ανήκει κάποιος, σε ποιες ε, πολιτικές πεπιθήσεις έχει. Και αυτό παρότι βασίζεται μόνο σε προσωπικά δεδομένα ή μεταδεδομένα έχει επιπτώσεις και σε αυτούς τους ε, τομείς. Τέλος, κάτι που είναι ανησυχητικό είναι μια νέα εξέλιξη στην Ευρώπη, τα βιομετρικά διαβατήρια. Σε πολλές χώρες τα βιομετρικά δεδομένα δεν ε, περιορίζονται μόνο στα διαβατήρια, αλλά συλλέγονται από εθνικές αρχές. Είναι λοιπόν απόλυτα δυνατό τα βιομετρικά αυτά δεδομένα να χρησιμοποιηθούν εναντίον προσώπων και να χρησιμοποιηθούν χωρίς να χρειάζεται συλλογή προσωπικών δεδομένων. Και τώρα ε, υπάρχουν αυτές οι βάσεις δεδομένων που θα συσταθούν βάσει αυτών των ε, βιομετρικών διαβατηρίων και Αυτές οι βάσεις, ε, έχετε και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διάφορα άλλα ζητήματα που θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εισαγωγή λοιπόν των βιομετρικών δεδομένων στα διαβατήρια έχει εφαρμογή και πέρα από τους ασυνοριακούς ε, ελέγχους. Πιστεύω λοιπόν πως υπάρχει απόλυτη ανάγκη επαγρύπνησης. Βέβαια εδώ υπάρχει και ένα ευρύτερο ερώτημα. Η δημιουργία της ε, μιας οχυρωμένης Ευρώπης, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα. Και αυτή είναι μία μόνο πτυχή του. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά. That's probably the video conference starting. Thank you for finishing. Ευχαριστώ λοιπόν που ολοκληρώσατε ενώ αναμένουμε την άνοιξη της βιντεοδιασκέψης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την συμβολή σας, ε, τις συστάσεις, ε, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμες προς τους σκιώδεις εισηγητές και σε μένα ως εισηγητή κατά τη σύνταξη της έκθεσης. Όλα αυτά θα τα αναρτήσουμε στο website ε, και οι συνάδελφοι που επιθυμούν μπορούν να τα δουν εκεί. Ευχαριστώ λοιπόν που ήσασταν σύντομοι και έτσι τελειώσαμε εγκαίρως την ε, συζήτηση. Ίσως να μην είμαστε ακόμα έτοιμοι για την βίντεο διάσκεψη. Λοιπόν, τώρα έχουμε την τηλεδιάσκεψη των ε, δικαστή Μπότζον ε, Πάντιτ. δεν ξέρω αν μας ακούει εντάξει μας ακούει ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα κύριε καθηγητά ευχαριστώ που είσαστε ανάμεσά μας um, well, this is a very complex problem legally speaking of course but primarily it is not a problem of the European law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 This would be my opening remarks. I am ready for any questions if you so want, sir. Thank you very much, uh, Judge Spanchik. And, uh... Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωσή σας. Έχουμε ένα άρθρο 8 το οποίο θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίασή μας. Υπάρχει λοιπόν επικάλυψη όπως καταλαβαίνετε.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 auch umgeht. Ähm, jetzt ist für mich nur die Frage in einer globalisierten Welt. Αναφερθήκατε στα εθνικά δικαιώματα. Εγώ όμως αναρωτιέμαι σε έναν κόσμο έτσι παγκοσμιοποιημένο τι κάνουμε σε περίπτωση παράκαμψης των εθνικών δικαιωμάτων όταν η μία μυστική υπηρεσία σε περίπτωση που εκείνη δεν ε, μπορεί να παρακολουθήσει κάποια συγκεκριμένα άτομα, απευθύνεται σε μια φιλική, φιλικά προσκύμενη άλλη εθνική μυστική υπηρεσία και τη ζητήσει να παρακολουθήσει τους ανθρώπους αυτούς εκ μέρους της. Τι προβλέπετε στην περίπτωση αυτή. Έπειτα, μια δεύτερη ερώτηση που ήδη υποβλήθηκε και όλας. Η αποθήκευση και μόνο των δεδομένων αποτελεί παραβίαση δικαιωμάτων προσωπικότητας ή παραβίαση καθιστά η ανάλυση και η χρήση αυτών των δεδομένων. Και τελευταία ερώτηση. Εσείς είχατε ποτέ τη δυνατότητα να ασχοληθείτε με μία υπόθεση αποθήκευσης δεδομένων για κάποιο χρονικό διάστημα. Thank you very much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 inwieweit für Sie das Speichern von Daten alleine schon eine Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte sein könnte. Κατά πόσο η αποθήκευση και μόνο αποτελεί παραβίαση δικαιωμάτων προσωπικότητας ε, κατά την άποψή σας ή θεωρείτε ότι μόνο η επεξεργασία των δεδομένων αυτών αποτελεί παραβίαση και όχι η απλή συλλογή τους. No, as I said, the storage alone is sufficient to constitute a violation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 Judge Sabanchik, I think you didn't hear Mr. Voss's first and... Νομίζω δεν ακούσατε την πρώτη και την τρίτη ερώτηση του κύριου Βόσα. The first question I didn't understand if you could repeat it. Yeah. Axel, if you could repeat the first question. And Die erste Frage beschäftigte sich mit dem. Η πρώτη ερώτησή μου αναφερόταν στην περίπτωση όπου, ε, όπως είπατε και εσείς, ε, είναι θέμα εθνικού δικαίου. Στα πλαίσια λοιπόν της παγκοσμιοποίησης και των ε, μυστικών υπηρεσιών και στα πλαίσια της ανταλλαγής δεδομένων υπάρχει περίπτωση κάτι που δεν επιτρέπεται να κάνει μια υπηρεσία, μια μυστική υπηρεσία να το αναθέσει στην άλλη. That's right. That's right. No, no, I understand I thought I, sort of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 Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Δικαστά για την παρουσίαση. Με καταθλίψατε, δεν φταίτε εσείς όμως, αλλά ε, οποιοδήποτε πολίτης ε, τα άκουγε όλα αυτά θα κατανοούσε ότι δεν έχει καμία νομική προστασία. Διότι ακόμα και αν υπήρχε θα ήταν αδύνατον να την ε, κατανοήσει. Αυτή η προστασία. ήμουν στο Λουξεμβούργο σε μια υπόθεση στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που με αφορούσε εγώ επέμεινα, αλλά αν είσαι ένας απλός πολίτης και θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματά σου, ε, ε, έχεις χάσει θεώρησα ιδιαίτερα σοκαριστικό ότι τα δικαστήρια δεν ασχολούνται διόλου με τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Και βλέπω ότι γνέφεται καταφατικά. Βλέπω όμως ότι δεν υπάρχει ουσιαστική νομική προστασία για τα δικαιώματα των πολιτών. Αυτό είναι το συμπέρασμά σας και εσάς.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 θα επανέλθουμε με καλά σε ό,τι φορά το χρόνο. Μία ερώτηση από την ομάδα των Παρσίνων, κύριε Δικαστά. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που δείξατε τόσο ανοιχτό πνεύμα σχετικά με την κατάσταση όταν αφορά την εφαρμογή της ε, Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδώ δεν μιλάμε μόνο στις με δραστηριότητες του NSA, αλλά και για το θέμα των, ε, των διαφόρων αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της Σύμβασης των, των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. θα μπορεί όλοι οι πολίτες να ε, βρίσκουν το δίκαιο τους, θα έλεγα. Υπήρχαν κάποιες υποθέσεις στο Στρασβούργο σχετικά με την ιδιωτικότητα, τα προσωπικά δεδομένα και το δικαστήριο είχε δηλώσει ότι μια έρευνα χωρίς ε, να υπάρχουν κάποιες υποψίες, κάποιες υπόνοιες, ε, δεν είναι συμβατή με το δικαίωμα της ιδιωτικότητας. Θα θέλω να μάθω πώς κρίνετε αυτήν την απόφαση, ποια είναι η θέση σας. Και ως δικαστής Πώς βλέπετε τη συλλογή και την ανάλυση των μεταδεδομένων σε σχέση με τα email. Είναι δικαιολογημένο σε σχέση με την ιδιωτικότητα ή περνάνε ακόμα και το θέμα της ιδιωτικότητας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 πιθανές ε, παραβιάσεις δεν είναι ορατές, θα πρέπει να αποδειχθούν από τον πολίτη. Πώς λοιπόν εγώ θα μπορούσα να πάω σε ένα δικαστήριο αν δεν έχω την δυνατότητα ως πολίτης βάσει κάποια σύμβασης τα δικαιώματά μου έχουν παραβιαστεί αν δεν υπάρχει διαφάνεια και οι κανόνες απορρίτου μου το απαγορεύουν. Νομίζω ότι είναι φαύλος κύκλος. Θα ήθελα να γνωρίζω την ερώτησή σας ως δικαστή. Τι γίνεται. Δεν μπορώ να τύχω δίκαιας δίκης σε ό,τι αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων μου. Υπάρχει τουλάχιστον δυνατότητα να προσφύγω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. in a situation where you cannot be certain, not positively certain, although it is probable, that you have been the victim of electronic surveillance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 το λόγο στους συναδέλφους αν έχουν ακόμα να θέσουν κάποια ερωτήματα στον δικαστή. Συνάδελφοι, έχουμε άλλες ερωτήσεις. Όχι μάλλον. Θα θέσω εγώ μία. Κύριε Δικαστά, εγώ θα ήθελα μάλλον στην επόμενη ε, μέρος της συνεδρίας να το συζητήσουμε, ώστε να έχω το σχόλιο και του καθηγητή ε, Κορφ. Μιας και προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο, Αναφέρομαι στο άρθρο 10 και 8. Είναι περισσότερο φιλοσοφικό το ερώτημα σε σχέση με το γεγονός ότι το δικαστήριο του Στρασβούργου είναι η τελευταία επιλογή. Επομένως, όταν το εθνικό νομικό πλαίσιο δεν είναι επαρκές, αναζητείται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το δικαστήριο του Στρασβούργου. Ε, στην επόμενη μέρος της συνεδρίασης θα εξετάσουμε μια υπόθεση ε, προσφυγής επί βάση του άρθρου 8. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι η εξή. Πώς βλέπετε το θέμα αυτό εσείς από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Γιατί όλο και περισσότερο στον Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη στο εθνικό επίπεδο και αυτό είναι ένα έλλειμμα όχι μόνο δικαστικό αλλά και πολιτικό. Τίθεται το, το θέμα της του κόστους της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θέλω να γνωρίζω τη δικιά σας θέση. Επίσης, έχουμε την, μια, μια κατάσταση στην οποία δημοσιογράφοι προσπαθούν να υπονομεύσουν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Δεν το υποστηρίζουν, ενώ οι πολίτες προσφεύγουν σε αυτό και αυτό είναι μάλλον παράδοξο. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας από αυτού, από αυτής της κατάστασης. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει έλλειμμα όσον αφορά την εθνική νομολογία. Θέτω αυτό το ερώτημα, θα ήθελα να γνωρίζω την άποψη και των συναδέλφων, αλλά πρώτα απ' όλα τη δική σας. Domestic remedies. Uh, in the UK. Um, so, for example, as Mr. Albrecht said, if you want a domestic remedy um, in a member state like the UK, it's actually very difficult. You're not going to get legal aid. You're not. Η κατάσταση σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει δωρεάν νομική βοήθεια. Επομένως δύσκολα μπορεί κανείς να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Η... Το θέμα του υπόθεση που θα εξετάσουμε αργότερα αφορά στην εξέβρεση πόρων από μεγάλο αριθμό οργανώσεων, αλλά ξαναγυρνώντας το ζήτημα της παρακολούθησης, είναι πολύ δύσκολο για έναν πολίτη ατομικά να προσφύγει κατά αυτής της παρακολούθησης. Το ερώτημά μου λοιπόν έχει σχέση με την εικόνα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που φαίνεται να έχει την εικόνα ε, του, του, του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Ενώ υπάρχουν και ορισμένε φωνέ που έχουν ζητήσει την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΣΔΑ και κατ' επέκταση από το δικαστήριο. the European Court of Human Rights and of the Convention that the subsidiary role of the European Court comes into play only after the domestic remedies have been exhausted. But to take a more cynical view of that, if you want, well, it's not really cynical, but it's a practical view, uh,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 Thank um, Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Δικαστά, και για την παρουσίασή σας. Το εκτιμούμε αυτό. Okay, and now we go... Ωραία και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρίτο μιλητή στο πάνελ αυτό. Okay, and this is the, um, this is the third session. Περνάμε λοιπόν στον τρίτο μιλήτη, ο οποίο θα μα μιλήσει για το δικαίωμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Είναι ο καθηγητής Ντόε Κόρφ, καθηγητή διεθνού δικαίου στο London Metropolitan University στο Λονδίνο. Ειδικεύεται σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο καθηγητής Κόρφ είναι γνωστό σε πολλού από εμά, και θα μα μιλήσει για την πτυχή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε το λόγο, κύριε Κόρφ. Ναι, ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή για την πρόσκληση σε αυτή την εξαιρετικά σημαντική συνεδρίασή της. Όπως αναφέρατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, στις προηγούμενες ακροάσεις είχατε ασχοληθεί περισσότερο με τα πολιτικά και τα τεχνικά ζητήματα, αλλά πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε και τον νομική πτυχή του θέματος. Ελπίζω να σας βοηθήσω λίγο ως προς αυτές τις πτυχές. Με την ιδιότητά μου ως δικαστής μπορώ... Ένας δικαστής μάλλον μπορεί να μας εξηγήσει καλύτερα την ΕΣΔΑ από ότι εγώ. Τώρα θέμα, στο, θέμα αυτό που αναφέρθηκε και πριν για το ζήτημα της ε, έσχατης προσφυγής. Υπάρχει μια πρόσφατη νομολογία του Δικαστήριο του Στρασβούργου ότι όταν δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης ενδικών μέσων τότε δεν τίθεται καν το θέμα της ε, εξάντλησή τους. Μου εξήγησαν ότι για να γίνω αγαπητός από αυτήν την επιτροπή θα πρέπει να τηρήσω το όριο των 10 λεπτών. Θα το προσπαθήσω. Αυτά τα λέμε πριν στους ομιλητές, λέει ο πρόεδρος. αλλά δυστυχώ οι διαφάνειες που προβάλλονται είναι η μακρά εκδοχή. Είναι μια παρουσίαση ενός υπομνήματος που κατέρτισα τον Αύγουστο. που αναφέρεται στην παρακολούθηση, θα έλεγα ότι μάλλον είναι μια πιο ακτιβιστική προσέγγιση, μια προσέγγιση περισσότερο κάποιου που ασκεί μια εκστρατεία πίεση. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να εστιάσω στα θέματα που αφορούν την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ περισσότερο και επίση για να μην επαναλάβω και αυτά που ήδη ακούστηκαν. Επίσης να επισημανώ ότι αυτό το έγγραφο είναι προσχέδιο, δεν είναι τελειώσει. Θα αναφερθώ λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύει την, τα προσωπικά δεδομένα και πώς ενσωματώνει τις ε, τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Το πρωταρχικό ζήτημα σε σχέση με το ε, εθνικό δίκαιο έχει σχέση με την σχέση μεταξύ της εθνικής ασφάλειας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Υπάρχει ήδη μεγάλη νομολογία, εκτενής νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Θα ήθελα κυρίως να υφιστήσω την προσοχή σας στην προσφυγή βέβαια και Σαβάρη εναντίον της Γερμανίας. Εξετάζοντας αυτή την απόφαση είναι αρκετά εύκολο να εξάγει κανεί ποιε θα πρέπει να είναι οι αρχές, τις οποίες θα πρέπει να σέβονται τα κράτη-μέλη όταν ασκούν δραστηριότητε παρακολούθηση, ποιε αρχέ κύπτουν από την ΕΣΔΑ. Και σας παραπέμπω κυρίως στην σελίδα 6, μια σελίδα η οποία περιληπτικά αναφέρει αυτές τις αρχές. Οι, τα κράτη υπέχουν θετικές υποχρεώσεις. Πρώτα απ' όλα να προστατεύουν τους ε, ε, τους πολίτες τους από την παρακολούθηση, καθώς επίσης και να προστατεύουν τους πολίτες τους από την παρακολούθηση από τρίτες χώρες. Αυτό είναι μια αρχή του διεθνούς δικαίου γενικότερα, η οποία προβλέπει ότι οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι υποχρεώσεις του κράτους από το διεθνές δίκαιο αφορούν και τους πολίτες και τους πολίτες ε, τρίτων χωρών. Επίσης, τα κράτη δεν έχουν τη δυνατότητα να ε, ασκούν ενέργειες οι οποίες θα ήταν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των πολιτών τους εναντίον πολιτών τρίτων χωρών ή στο έδαφος τρίτων χωρών. Χρειάζονται λοιπόν αυστηροί κανόνες για την παρακολούθηση, συγκεκριμένη νομική βάση για τον στόχο και για το χρονικό πλαίσιο. Ο κύριος Νίκλ Πίκλς μάλλον θα μας εξηγήσει καλύτερα την κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο με βάση την υπόθεση που θα μας παρουσιάσει. το ζήτημα της εξωεδαφικής εφαρμογής το ανέφερα ήδη. Πιστεύω ότι σε σχέση με την ΕΣΔΑ το ε, θέμα της ετεροδικίας πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στα ζητήματα ε, ε, προστασίας προσωπικών δεδομένων το δικαστήριο του Στρασβούργου έχει ήδη ασκήσει κριτική επικρίσεις σε σχέση με την γενικευμένη παρακολούθηση, την μαζική παρακολούθηση. Πιστεύω ότι και το δικαστήριο του Λεξεμβούργου θα ακολουθούσε την ίδια τακτική σε περίπτωση που ένα κράτος επιχειρηματολογούσε με βάση την ε, εθνική του ασφάλεια για να δικαιολογήσει τη μαζική παρακολούθηση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επαναλάβω ποιε είναι οι γενικέ αρχέ τη προστασία ε, προσωπικών δεδομένων. Αυτές, αυτή η επεξεργασία πρέπει να γίνεται με τρόπο δίκαιο, με τρόπο διαφανή. Θα πρέπει να είναι σαφέ ο σκοπό τη επεξεργασία. Ε, τα υποκείμενα τη επεξεργασία έχουν δικαιώματα κτλ. Αυτά είναι γνωστά. Αλλά πρέπει να παρατηρήσω ότι η παρακολούθηση την οποία ε, άσκησε το Ηνωμένο Βασίλειο και από ό,τι φαίνεται και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εντελώ πλήρω 100% παραβίαση της θεμελιώδους νομοθεσίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της θεμελιώδους νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι ξεκάθαρο και νομίζω στην επόμενη διαφάνεια θα γίνει ακόμα πιο σαφές. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη έχει διεξαχθεί σε σχέση με τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων για την αποθήκευση δεδομένων. Είναι επικίνδυνη αυτή η αποθήκευση δεδομένων για μακρά χρονικά διαστήματα γιατί μπορεί να διευκολύνει την μαζική παρακολούθηση και την μαζική εξόριξη δεδομένων. Το θέμα του data mining λοιπόν, της ε, εξόριξης δεδομένων της εφαρμογής αλγοριθμών τεχνητής, νοημοθεσ... Ε, νοημοσύνης, για την βελτίωση των αλγορίθμων αναζήτησης με βάση τις λέξεις κλειδιά. Όλα αυτά τελικά οδηγούν στη δημιουργία ενός προφίλ. Η δημιουργία προφίλ για, έναν, για κάποιον χρήστη, για κάποιον άνθρωπο είναι από τη φύση της επικίνδυνη όταν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το προφίλ του τρομοκράτη είναι αναπόφευκτο ότι θα δημιουργήσουμε πάρα πολλές, ε, πολλούς ψεύτικους συναγερμούς. Θα, θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου το σύστημα θα μας ε, υποδείξει κάποιον ως τρομοκράτη χωρίς αυτό να ισχύει. Και αυτό θα καταστρέψει προφανώς τη ζωή πολλών πολιτών πέρα από τα ζητήματα προστασίας δεδομένων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γενικότερα τίθενται. Έχω εδώ ένα παράδειγμα που αναφέρεται στη νομοθεσία, μια περιοριστική νομοθεσία και η οποία σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα για να σας δείξω ότι αυτό είναι εφικτό. Τι έχουμε εδώ, μια, ένα σαφή ορισμό του σκοπού της επεξεργασίας. Ποιο, με, βάση ποιο σκοπό συλλέγονται αυτά τα δεδομένα. Και θα επανέλθω μετά στο ζήτημα της εξαίρεσης με βάση τις την εθνική ασφάλεια. Το ζήτημα θα πρέπει να είναι, το, το, η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να έχει σαφή στόχο. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να έχει επιλεγεί με βάση αποδείξεις ή ενδείξεις. Επαρκούν και οι ενδείξεις, αλλά θα πρέπει αυτές οι ενδείξεις να ήταν σαφείς, τόσο σαφείς, έτσι ώστε να οδηγούν σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα άτομα. Δεν είναι αποδεικτή μια μαζική παρακολούθηση οποιοδήποτε δυνητικά στο μέλλον θα μπορούσε να ε, προχωρήσει σε έκνομες πράξεις. Και τώρα για να επιβεβαιώσω αυτά που είπε και ο Μάρτιν σε σχέση με τις αρχές που εφαρμόζονται στην Ευρώπη είναι ακριβώς οι ίδιες με εκείνες που προβλέπεται στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Δηλαδή ότι χρειάζεται να είναι σαφής σαφές το, το δίκαιο, να υπάρχει ασφάλεια δικαίου, να είναι δημόσιο, δεν είναι δυνατόν αυτές οι αποφάσεις να λαμβάνονται από μυστικά δικαστήρια, θα πρέπει επίσης να γίνεται σεβαστή η αναλογικότητα. Οι διεθνείς λοιπόν υποχρεώσεις, οι διεθνείς ρήτρε και οι ευρωπαϊκές ρήτρε είναι ίδιες. Ε, υπάρχει επίσης η ισότητα των πολιτών και των, μη, ε, των υπηκών και των μη υπηκών μιας χώρας. Με τον ίδιο τρόπο προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα ενό προσώπου ανεξαρτήτως από το εάν είναι πολίτη ή όχι μιας χώρας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι λοιπόν μέρος του ICCPR και θεωρώ ότι μια διακρατική προσφυγή εναντίον τους θα ήταν σκόπιμη, θα πολύ χρήσιμη και θα ε, βελτιώσει και την ε, προστασία του ICCPR. Παρεπιπτόντος, όταν κάποια χώρα ασκεί δραστηριότητε παρακολούθηση στο έδαφος άλλης χώρας, αυτό παραβιάζει και το δικαίωμα της κυριαρχίας. Κάτι που έχει παραδεχτεί και σε απόφαση το 1927 το ε, διεθνέ Δικαστήριο, το Δικαστήριο Διεθνούς Δικαίου της Χάγης. Επομένως, εδώ τα κράτη που επιδίδονται σε τέτοιες διαστριότητε παραβιάζουν γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου. Και ένα πιο συγκεκριμένο ε, ζήτημα. Υπάρχει μια πρόταση για ένα νέο προαιρετικό πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ, η οποία το οποίο σε περίπτωση που συνευθεί θα μπορούσε να νομιμοποιήσει αυτή την διασυνοριακή συλλογή δεδομένων από τις υπηρεσίες ασφαλείας. Πρέπει να, γίνει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και σας ζητώ και εσείς να το πράξετε για να σταματήσουμε την υιοθέτηση αυτού του πρωτοκόλλου. Και τώρα έρχομαι στο θέμα που κυρίως με ενδιαφέρει. Και αυτό είναι το θέμα της εξαίρεσης εθνικής ασφάλειας στις συνθήκες και πιστεύω πως αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Αν διαβάσουμε το άρθρο 4.2 αναφέρεται ότι η εθνική ασφάλεια είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι δηλαδή αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών, καμία αρμοδιότητα διαφορετικού συμβαλωμένου μέρου. Το δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα. Αυτή είναι και η νομική θέση. Και πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε όλοι αυτό. Τώρα, το πρώτο ζήτημα που προκύπτει είναι το εξή. Υπάρχει ένα μεγάλο εύρο αρμοδιοτήτων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε ζητήματα όπω η εσωτερική ασφάλεια και εδώ εννοώ την εσωτερική ασφάλεια τη Ένωση. Την κοινή, πολιτική, την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, η οποία ασχολείται και με πολλά θέματα διεθνούς δικαίου και επίσης υπάρχουν αρμοδιότητες ε, σε σχέση με τρομοκρατία και σοβαρά εγκλήματα ε, στο Συμβούλιο Υποθέσεων. Όλα αυτά είναι, είναι πτυχές που δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε από το ζήτημα της εσωτερικής ασφάλειας. Υπάρχει γενική νομοθεσία των συνθήκων όπου αναφέρεται ότι τα κράτη δεν επιτρέπεται να ε, δρούν με τρόπο που να υπονομεύει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συνθήκη. Τι σημαίνει αυτό, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να, ε, για θέματα εθνικής ασφαλείας ε, να πράττει με τρόπο που υπονομεύει αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, την διεθνή εξωτερική ασφάλεια και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος. Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι άλλες χώρες εξάλλου έχουν καθήκον να ε, υπηρετούν τα συμφέροντα της εσωτερικής ε, ασφάλειας ε, με τρόπο όμως που να είναι σύμφωνος με αυτά που προβλέπουν οι συνθήκες και αυτό απαγορεύει οτιδήποτε, οποιαδήποτε δράση υπονομεύει και παραβιάζει τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό είναι το ένα λοιπόν ζήτημα, αρμοδιότητα της Επιτροπής και γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμοδιότητα για έλεγχο εάν το Ιωνωμένο Βασίλειο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συνθήκες. Και επίσης υπάρχει και το θεμελιώδες ερώτημα του τι καθιστά εθνική ασφάλεια. Έχουμε δει, ιδιαίτερα στις Ηνωμένε Πολιτείε με το ΦΙΣΑ, ε, ότι υπάρχει ένας ε, ευρύτατος ε, ορισμός του τι συνιστά εθνική ασφάλεια για εκείνους. Και σύμφωνα με αυτό μπορούν να συλλέξουν οτιδήποτε θα μπορούσε να σχετίζεται με τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ ή με την εσωτερική της ασφάλεια. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει βιομηχανική κατασκοπία, απλή κατασκοπία, ε, παρακολούθηση μη βίων πολιτικών ομάδων, όπως για παράδειγμα η Big Brother Watch που έχουμε μαζί μας, ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις για δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, για παράδειγμα το ε, αυτά λοιπόν ε, για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Τώρα, ορισμός του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός στο, ε, στη Βρετανική νομοθεσία και παλαιότερα ορισμός της εθνικής ασφαλής ήταν τον, οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο την ε, ε εθνική ασφάλεια, πανδημίες, ε, γενικότερες απειλές και το το Ηνωμένο Βασίλειο επίση ε, να πω ότι απέρριψε στο δικαστήριο μία υπόθεση δωροδοκίας ε, για το λόγο ότι έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Έχουν προκύψει ορισμένοι ενδιαφέροντες ορισμοί με βάση λοιπόν την νομολογία του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την εθνική ασφάλεια. Επίση, σα αναφερθούμε στι αρχέ του Johannesburg, οι οποίε έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 και τις οποίες έχουν εγκρίνει ε, μια, ένας αριθμός διεθνών οργανισμών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας από αυτούς που αναφέρονται σε ορισμούς εθνικής ασφάλειας. Η εθνική ασφάλεια λοιπόν, ε, σύμφωνα με αυτό, στόχο έχει να ε, προστατεύσει ένα κράτος από εξωτερική βία, εξωτερική άσκηση βίας και δεν είναι ενόμιμη η χρήση για περιπτώσεις απόκρυψης πληροφοριών, απόκτηση διπλωματικού πλεονεκτήματος ή εμπορικών επιχειρησιακών πλεονεκτημάτων. Από τότε που ο ορισμός, ο πόρος Εθνική Ασφάλεια, άρχισε να χρησιμοποιείται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει μετατραπεί σε μια νομική έννοια στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, παρότι δεν έχει μεγάλη δικαιοδοσία για τις επράξεις των κρατών μελών, έχει δικαίωμα ερμηνείας της νομοθεσίας αυτής ε, σχετικά με το κατά πόσο συμφωνεί με τις ε, συνθήκες. Αυτό είναι ο ευρύτερος ε, ορισμός. Τώρα θα ήθελα να περάσω στα σχόλιά μου για την ε, ευρωπαϊκή, για την ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Όπως βλέπετε και εδώ, οι αρμοδιότητες περιορίζονται σε θέματα εθνικής ασφαλείας έτσι όπως αυτή ορίζεται από το Διεθνές Δίκαιο. Ακόμα και αν οι πράξεις του Ηνωμένου Βασιλείου περιορίζονται σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας έτσι όπως το καταλαβαίνουμε από το δίκαιο, υπάρχει ακόμα το εκρεμές ζήτημα του αν οι πράξεις αυτές υπονομεύουν τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε κοινέ είτε μη κοινέ. Ε, οι αρμοδιότητε που σχετίζονται με την ασφάλεια, την καταπολέμηση τη τρομοκρατία ε, και των ε, σοβαρών εγκλημάτων. Και φυσικά σε περίπτωση που η Επιτροπή, το δικαστήριο μάθαινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ή κάποιο άλλο κράτος δεν περιοριζόταν σε ε, εσωτερική ασφάλεια, τότε δεν θα καλυπτόταν από την εξαίρεση του άρθρου αυτού. Και αυτές οι επιπλέον εξωτερικές ε, δραστηριότητες θα ε, υπόκειται στην αρμοδιότητά του λοιπόν. Όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή αυτή έχει την αρμοδιότητα ελέγχους για το αν οι Ηνωμένε Πολιτείες συμμορφώνονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ε, ασκούν στην επικράτειά της. Και φυσικά σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις ε, συμφωνίες για τα δεδομένα των επιβατών και τη συμφωνία ε, SWIFT. Και με, το, με, το, με τους ασφαλείς ελιμένες. Να σας πω ότι συμφωνώ και με τον συμπατριώτη μου, τον Πέτερ Χόστινγκ, για το ότι αντιμετωπίζουμε μια πολύ σημαντική πρόκληση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό σε μια εποχή όπου κινδυνεύουν τα βασικά μας δικαιώματα, βασικά μας κοινωνικά δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ζήτημα του Safe Harbor των ασφαλών ελιμένων είναι κάτι που θα εξετάσουμε διεξοδικά σε αυτή την Επιτροπή. Και η παρουσίασή σας θα ανέβει στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Να σας πω ότι η απουσία των μελών μας οφείλεται σε ε, λόγους. Λυπούνται πάρα πολύ που απουσιάζουν και θα ήθελαν να στείλουν ε, την εκτιμησή τους ε, για την ε, παρουσία σας. Τώρα, ο κύριος Γιάννα Άλμπρεχτ έχει πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, γιατί πιστεύω πως ασαφώς υπάρχει η παραβίαση του συμφώνου και του νομικού πλαισίου του. Η ερώτηση μου λοιπόν, όπως είπατε και εσείς ε, στην αρχή καθώς παρουσιάσατε τον τρόπο που μπορούν ε, τα, ε, οι πολίτες μεμονωμένα να αντιμετωπίσουν ε, με τέτοια παραβίαση, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν εάν υπάρχει ε, δυνατότητα για τα κράτη-μέλη, για τα θεσμικά όργανα να, να προσφύγουν στο δικαστήριο στο Στρασβούργο και αν ναι θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, εσείς θεωρείτε ότι για παράδειγμα στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχει ανάγκη πολιτικής ε, συζήτησης για τις ε, παραβιάσεις ε, του συμφώνου για τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα και για τον ε, τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν το σύμφωνο αυτό και τις συνθήκες και επίσης από άποψη σε διεθνούς δικαίου και διπλωματία. Σε ποιες είναι οι επιμέρους λεπτομέρειες. Θα θέλατε να απαντήσετε τώρα, λέει ο ή αργότερα. Ναι, θα ήθελα να σας απαντήσω όσον αφορά το δικαστήριο του Στρασβούργου που δεν μπορεί να ε, αλλάξει η νομοθεσία όπως μπορεί για παράδειγμα το συνταγματικό δικαστήριο στην Γερμανία δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Σε πολλές χώρε της Ευρώπης η νομοθεσία έχει αλλάξει ακριβώς εξαιτία του δικαστηρίου στο Στρασβούργο. Υπάρχει ένας μηχανισμός εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων του Στρασβούργου, ή μια επιτροπή υπουργών για παράδειγμα, και αυτό είναι μια βελτίωση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Εάν ε, διαπιστωθεί ότι υπάρχει παραβίαση του συμφώνου, τότε το κράτος μέλος που, κάνει την, που ε, κάνει την παραβίαση είναι υποχρεωμένο να λάβει μέτρα και να αλλάξει η νομοθεσία. Πιστεύω λοιπόν πως να υπάρχουν δυνατότητες μέσα στην Ευρώπη να διερευνηθούν κάποια ζητήματα. Τώρα ε, όσον αφορά την περίπτωση του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο. Δεν είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα από ότι στο Στρασβούργο. Δεν έχουμε επαρκής, ε, επαρκή ένδικα μέσα. Και σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, να πω ότι εδώ είναι προφανής η ανεπάρκεια του μηχανισμού εκεί, διότι δεν μπορούσε να σταματήσει την παραβίαση του συμφώνου. Εάν υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής άμεσα στο Στρασβούργο και το Στρασβούργο μπορούσε να εκδώσει μια απόφαση ή για παράδειγμα να δοθεί εντολή για διερεύνηση σύμφωνα με το άρθρο 52, αυτό θα ήταν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο ελπίζω το Συμβούλιο της Ευρώπης να ασκήσει την εξουσία που έχει σχετικά με αυτόν τον τομέα. Πιστεύω πως ε, αυτό θα δημιουργούσε ένα πολύ καλό προηγούμενο όσον αφορά τη δυνατότητα που θα έχει το δικαστήριο στο Στρασβούργο να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Ένα... Είναι προτιμότερο φυσικά να διαβάσουμε το κείμενο του συμφώνου όπου αναφέρονται τα απτά στοιχεία όπου αναφέρεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέσα στο κείμενο. Επίσης, ε, συμφωνώ απόλυτα με τον ε, καθηγητή Σάινιν στην παρουσίασή του. Πιστεύω πως ε, αυτό που χρειάζεται καταρχάς είναι να αναζητήσουμε τις ε, σωστές λύσεις. Ε, κάτι άλλο τώρα. Πριν από μερικά χρόνια διερεύνησα τις υποθέσεις προσφυγής κατά της Τουρκίας για, τον, για τα βασανιστήρια και υπήρχε μία προσφυγή 5 ή 7 κρατών. Θα ήταν καλύτερο να είναι ένα το κράτος που προσφεύγει και τα υπόλοιπα να έχουν δεύτερο ρόλο παρά να έχουμε τρία, τέσσερα, πέντε διαφορετικά κράτη, υπουργεία, αρμόδια υπουργεία που θα προσφεύγουν. Αυτό Ισχύει και για την ε, περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, μια, ένα έτοιμα έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 52 και διερεύνηση δυνατοτή, δυνατότητας ε, ανάληψης δράσης από το δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Κυρία Ζίπελ. Όχι, με συγχωρείς. Γιάννη, ήθελες να ρωτήσεις κάτι συμπληρωματικό. Ναι, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το χρόνο της κυρίας ε, Ζίπελ, αλλά να πω ότι Αυτό που έχω στο μυαλό μου συνδέεται με το διεθνές δίκαιο και καθώς είστε ειδικό στο διεθνές δίκαιο, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν εσάς. Προσωπικά θεωρώ πως πρέπει να ασχοληθούμε και με τις ε, επιθέσεις κατά της εθνικής κυριαρχίας των ε, κρατών. Σαφώς ε, διαπιστώθηκε μία επίθεση του Ηνωμένου Βασιλείου στην εθνική κυριαρχία του Βελγίου. Και ταυτόχρονα παρόμοιες επιθέσεις διεξάγονται από τις Ηνωμένε Πολιτείε σε άλλα κράτη-μέλη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ παρατηρούμε την ε, διάβρωση της εθνικής κυριαρχίας και δεν μπορώ να σκεφτώ κάποια άλλη περίπτωση ο, με τόσο μεγάλη μεγάλης κλίμακας επίθεση σε εθνική κυριαρχία, η οποία να έχει αντιμετωπιστεί με, τέτοιο, με τόσο αδύναμο τρόπο. Ε, τώρα, όταν ε, κάνουμε λίγο για διεθνές δίκαιο, σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δρούν με τον τρόπο που ε, δρούν σε αυτή την περίπτωση, τότε αυτές οι παραβιάσεις θα γίνονται αποδεκτές και το μελλοντικό διεθνές δίκαιο θα βασιστεί στις ε, περιπτώσεις αυτών των χωρών που παραβιάζουν το σύμφωνο. Εσείς, ποιες είναι οι επιπτώσεις που θεωρείτε ότι θα έχουν αυτές οι πρακτικές ε, στην ε, νομοθεσία που έχουμε πασχίσει να δημιουργήσουμε τόσα χρόνια. Μάλιστα, υπάρχει περίπτωση να προσφύγουμε στο δικαστήριο της Χάγης. Βέβαια, γι' αυτό χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη και των ε, δύο ε, αντιδίκων. Εάν και τα δύο κράτη-μέλη αντιτίθενται σε αυτό, τότε δεν θα δημιουργηθεί διεθνές εθνικό δίκαιο. Ε, σε περίπτωση που τα κράτη-μέλη δηλώσουν ε, ρητά ότι δεν εγκρίνουν αυτές, ε, αυτήν την διαδικασία. Τι γίνεται όμως, ρωτάει ο κύριος Άλμπρεχτ, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Να σας πω, πριν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι μυστικές υπηρεσίες έκαναν ό,τι ήθελαν. Από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά όμως, και μετά από πολλούς κοινοβουλευτικές επιτροπές ελέγχου, οι μυστικές υπηρεσίες δεν έχουν έρθει έχουν μπει εντό του πλαισίου του κράτου σε δικαίου. Στέκονται έτσι κι αλλιώς στο περιθώριο και δρούν σε αυτό το περιθώριο. Και αυτές οι διαδικασίες παρακολούθησης έχουν αρχίσει να παρισφρίουν σε πολλούς τομείς της, της ιδιωτικής ζωής. Και αυτός είναι ο κίνδυνος που έχει δημιουργηθεί από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας όλες οι συνθήκες, όλες οι διεθνείς συμφωνίες που έχουμε, που είναι και η βάση της ενομοθεσίας, όλη αυτή η συνεργασία λοιπόν ανάμεσα στις εμιστικές υπηρεσίες είναι κάτι που πρέπει να αναθεωρηθεί. Υπάρχουν οι συνθήκες, ε, συνθήκες του ΝΑΤΟ για παράδειγμα, τις οποίες δεν έχω δει ποτέ διότι είναι απόρριτε. Υπάρχουν συνθήκες ε, και νομίζω και ανάμεσα στη Γερμανία και σε κάποια άλλα κράτη ε, για τι οποίε κανείς δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Πιστεύω πως ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν απόρριτε συνθήκες. Όλα θα έπρεπε να βασίζονται σε ξεκάθαρου σε διάφανους, δημοκρατικούς κανόνες οι οποίοι θα έχουν εγκριθεί δημοκρατικά από κοινοβούλια. Πιστεύω πως για πάρα πολύ καιρό έχουμε ζήσει σε μια κοινωνία που κανείς δεν βάζει κάποια όρια. Κυρία Ζήπελ, ευχαριστώ πολύ. Αυτή η συζήτηση άρχισε με αφορμή την μαζική συλλογή δεδομένων από τις Ηνωμένε Πολιτείες και Έχουμε διαπιστώσει σήμερα ότι αυτή, αυτή η πρακτική παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες και τα, κράτη, και τα κράτη δεν αντιδρούν σε αυτή την παραβίαση. Αναφέρθηκε επίσης ότι τουλάχιστον ε, στα χαρτιά η Ευρώπη έχει καλύτερες συνθήκες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, είναι όντω οι καλύτερες συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη ή είναι μόνο στα χαρτιά. Έπειτα, ο ορισμός τη εθνικής ασφάλειας στις συνθήκες ως αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Είναι κάτι που με έκανε πάντα να απορώ, διότι η εθνική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και η μάχη κατά της τρομοκρατίας είναι επίσης ε, λοιπόν θέμα εθνικής ε, ασφάλειας. Όμως οι, εθνικές, οι εθνικές αμυστικές υπηρεσίες συνεργάζονται και ανταλλάσσουν δεδομένα. Θα ήθελα να ακούσω λοιπόν την τοποθέτησή σας ε, για αυτό το θέμα. Εάν υπάρχει μια ευρωπαϊκή διάσταση στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και τέλος, πράγματι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν επιτροπές ελέγχου, υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι όμως δεν λειτουργούν πάντοτε όπως θα έπρεπε. Όμως, όπου υπάρχει ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, έχω εγώ τη δυνατότητα, έχει ένα κράτος μέλος τη δυνατότητα να ζητήσει να τηρηθούν οι κανόνες της διαφάνειας και της αναλογικότητας ε, στην ε, δράση των μυστικών υπηρεσιών και τη βελτίωσή τους. Να προσθέσω κι εγώ κάτι, λέει ο Πρόεδρος. Και μετά θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Μία ερώτηση και μετά να κάνετε μία τελευταία, με τελευταία απάντηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την εξαίρεση εθνικής ασφάλειας και να μιλήσετε επίσης για την υπόθεση Belgacom. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι είχαμε αυτό το ad hoc, ε, ad hoc ακρόαση με την Belgacom Εάν ε, δεν έχετε κάποια γενικότερη άποψη για το ζήτημα, η συνθήκη αναφέρει ότι υπάρχουν αυτές εξαιρέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Πώς ε, μπορείτε να διευθυντήσετε ένα παρόμοιο ζήτημα. Υπάρχουν κάποιες θέσεις αναφορικά με τις ε, υπηρεσίες ασφάλειας, ε, πληροφοριών και τι γίνεται αν υπάρχουν ισχυρισμοί από κάποια κράτη-μέλη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου υπάρχουν διάφοροι ισχυρισμοί βάσιμοι και οι δύο προέρχονται από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος πολίτης πώς μπορεί να κατανοήσει κάτι τέτοιο. Ότι υπάρχει εμπλοκή της Europol, θέματα εσωτερικής ασφάλειας. Äh, Θα ήθελα καταρχάς να προσπαθήσω να απαντήσω, να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας, κύριε Ζήπελε. Πριν από ένα μήνα υπόθηκε από τους Αμερικανούς ε, το εξής. Γιατί είμαστε πάντα οι κακοί, ενώ εσείς δεν είστε καλύτεροι από εμά. Αναρωτήθηκα λοιπόν γιατί το είπαν αυτό. Ήξεραν κάτι που εμείς δεν ξέραμε, προφανώς και ναι. Και αυτό το θεώρησα πολύ ενδιαφέρον. Όντως, είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη τα πράγματα είναι καλύτερα στα χαρτιά. Υπάρχει το, η Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δεν υπάρχει καμία εξαίρεση σε θέματα εθνικής ε, ασφάλειας. Φυσικά, αναρωτιέται κανείς ε, ναι, τι συμβαίνει όταν ε, δεν τηρούνται αυτές οι συμβάσεις. Ποιος έχει την αρμοδιότητα, το δικαστήριο του ε, κράτους ε, μέλους ή το δικαστή, η Σύμβαση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το Στρασβούργο, ποιος έχει την αρμοδιότητα. Η αρχή είναι σαφής ε, για μένα. Και οι δικαστές πιστεύω πως δεν θα έπρεπε να έχουν πρόβλημα να αποφασίσουν ποιος έχει αρμοδιότητα σε μια τέτοια υπόθεση. Τώρα στις οι Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχει η πρώτη τροπολογία, η οποία, σύμφωνα με την οποία ε, η οποία μάλλον θεωρείται ένα πολύ μεγάλο λάθος του αμερικανικού συστήματος. Τώρα όμως, τι γίνεται στην πράξη. Πιστεύω πως ε, τώρα που ξέρουμε τι έχει συμβεί, έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να δούμε τα γεγονότα με γυμνόφθαλμό και να τα εξετάσουμε. Τώρα, ο πρόεδρος ρώτησε πώς μπορούμε λοιπόν να μάθουμε αυτές τις ε, πληροφορίες. Και η κυρία Ζήπελε ρώτησε κάτι παρόμοιο επίσης. τρομοκρατία. υπάρχουν ευρωπαϊκές αρμοδιότητες για την τρομοκρατία. Δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μείνει εκτός επειδή είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας και το δικαστήριο στο Λουξεμβουργό έχει αποφανθεί γι' αυτό ε, σχετικά με το πώς μπορεί να ενεργήσει ένα κράτος ε, μέλος, τι ε, μπορεί να κάνει σε θέματα εθνικής ασφάλειας, σε θέματα τρομοκρατίας και ποιες είναι οι ευρωπαϊκές αρμοδιότητες και πώς αυτές σε συνδυάζονται. Ε, όμως ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο είναι το μόνο αρμόδιο για επίλυση θεμάτων ευρωπαϊκής ή εθνικής αρμοδιότητας. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι έχει αρμοδιότητες ε, και ο διαχωρισμός είναι ε, καθαρά νομικό θέμα το οποίο θα εξετάσει και για το οποίο θα αποφανθεί το δικαστήριο. Τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημα του Πρόεδρου. Τι μπορούμε να κάνουμε όταν ζητείτε εξαίρεση με βάση την εθνική ασφάλεια από ένα κράτος μέλος, το οποίο θα επηρεάσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα πολιτών ενός άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει την Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση, θα πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση σε αυτό. Εάν μιλούμε για μια για την σύγχρονη κοινωνία στην οποία υπάρχουν όλες αυτές οι απειλές τρομοκρατίας που έχουν οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρεί ότι πρέπει να συνεργαστεί για την προστασία των πολιτών της. Και ταυτόχρονα ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της από την υπερβολική κρατική ε, νομοθεσία αντιτρομοκρατίας τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να λάβει θέση. Δεν εννοώ να υπαγορεύσει τις λεπτομέρειες, αλλά τις βασικές αρχές. Η εθνική νομοθεσία εθνικής ασφάλειας θα μπορούσε να τεθεί υπό τον, ε, να εξεταστεί από τον στο επίπεδο του Ευρωπαϊκή Ένωση και στο επίπεδο του, Ευρωπαϊκού, του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Ε, τη στιγμή που τα κράτη λένε ότι σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο πρέπει όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε για να αντιμετωπίζουμε τι απειλέ. Πώ μπορούν να το λένε αυτό από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά να λένε ότι ναι, ε, ε, δεν θέλω κανεί να ασκήσει κριτική στον τρόπο με τον οποίο ασχολούνται και ασχολούμαι με τι εσωτερικέ μου υποθέσει. Σα ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω και του τρει ομιλητέ. και νομίζω ότι τώρα μπορεί να αλλάξει το πάνελ και να συνεχίσουμε την επόμενη σύνοδο.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 Συνάδελφοι, προχωράμε στο δεύτερο πάνελ, στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασής μας. Όπως είπα στην αρχή, θα εστιάσουμε στις εκκρεμείς ε, δικαστικές υποθέσεις από τότε που ε, διαπιστώθηκαν οι κατηγορίες για μαζική παρακολούθηση. Θα ασχοληθούμε με δύο συγκεκριμένες υποθέσεις και προτείνω καταρχάς να ακούσουμε τους τρεις ομιλητές και μετά να προχωρήσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Θα αρχίσουμε με την υπόθεση στο Παρίσι ε, κατά γνώστου. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Ντομινίκη Ζιμπέρ, αντιπρόεδρο της ε, Λίγας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα ζητήματα σχέση με αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, πρώτη σκέψη είναι οι σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και την ε, και τα δικαιώματα. Δεν θέλαμε λοιπόν λόγω της ε, να, να παραπέσουμε σε ένα από τα δύο θέματα, να δώσουμε μεγαλύτερη βάση στο ένα από τα δύο θέματα. Δηλαδή να εκδικαστούν κάποιες υποθέσεις ε, με βάση την αρχή ότι η δικαιοσύνη περισχύει της ελευθερίας. Και κάτι ακόμα, είπαμε ότι υπάρχει η <clears throat> τέταρτη τέταρτο άρθρο του συντάγματος του ε, για τους πολίτες και είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να σημαίνει για τα άλλες υποθέσεις και ότι και όχι επειδή υπάρχει κάποιο σφάλμα ουδήποτε θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε άλλες περιπτώσεις με άλλα λόγια επειδή είναι ε, παράνομο στα κράτη στις ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι νόμιμο και αλλού το τρίτο αφορά την έννοια του απορρίτου. Διαπιστώσαμε ότι ακόμα και όταν οι Αμερικανικές αρχές δηλώνουν ότι το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο εποπτεύουν αυτά τα θέματα των ελέγχων των επικοινωνιών ή άλλων, όλα αυτά παραμένουν στο πλαίσιο του απορρίτου. Αλλά το απορρίτο, το απορρίτο δεν είναι κάτι δημοκρατικό, δεν μπορεί να ελέγχεται από τον πολίτη και να υπενθυμίσω την ε, το Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Γαλλία, όπου με την υπόθεση τρέφου αυτό που είχε απαντηθεί στου δικηγόρου που ζητούσαν τη δημοσίευση των ε, στοιχείων που ζητούσαν ε, το δικαστήριο, είχαν πει ότι δεν πρόκειται να καρδεθούν. Και τώρα, Κάτι ακόμα, το θέμα της ασφάλειας. Η εσωτερική ασφάλεια κατέστη τώρα, μάλλον επεκτάθηκε και αφορά το σύνολο της ασφάλειας. Η εσωτερική ασφάλεια αφορά και την εξωτερική ασφάλεια. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να συνδέσουμε όλες αυτές τις ερωτήσεις, όλα αυτά τα ζητήματα ελέγχου των συνόρων και ελέγχου των πολιτών σε αυτά τα οποία εμπίπτουν στον όρο ε, οχυρό. Ο όρος οχυρός με στο να ε, θεωρείς ότι είναι τραγικός αυτός ο όρος, είναι ο ίδιος όρος με τη Λαμπεντούζα. Όπως ε, είπε ο πρόεδρος, θα αναφερθούμε τώρα στην ε, υπόθεση που έχουμε καταθέσει ενώπιον του Δικαστήριου των Παρισίων, την Ευρωπαϊκή, την, τον 11 Ιουνίου 2013 αναθέσαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μάλλον στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μια αγωγή κατάχη για τα θέματα που αφορούν την υπόθεση Snowden, τόσο για το κοινωνικό δέσμα που οδηγεί στην ε, απόπειρα των ε, ε, επιρροής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταθέσαμε λοιπόν κάποια στοιχεία για την παραβίαση της συλλογής δεδομένων με ε, απόπειρα κατά της ε, ζωής ε, και την καταγραφή γράφων απόπειρα κατά της προσωπικής ελευθερίας. Και η υπόθεση Νόιντον μας έκανε να αποκαλύψουμε το πρόγραμμα των Αμερικανών που φωνάζεται Prison. Η καταπαλήμψη της τρομοκρατίας και αυτή η, αυτός ο έλεγχος των ιδιωτικών στοιχείων ε, επέτρεψε στην NSA και την FBI να συλλέξουν ε, ε, πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Αυτό το σύστημα λοιπόν το οποίο οδήγησε σε έλεγχο 500 εκατομμυρίων στοιχείων αναμίνα επέτρεψε όχι μόνο να συλλέξουν στοιχεία για την προέλευση αλλά και για τον παραλείπτει αυτά των μηνυμάτων. Αυτή λοιπόν η εισβολή, η ανεξέλεγκτη στην ιδιωτική ζωή αποτελεί κίνδυνο για τις ατομικές ελευθερίες που θα πρέπει να διαγραφεί για να μην θέσουμε να αμφιβόλο το κράτος δικαίου. Οι LDA και FDA ανέθεσαν στην ε, γαλλική δικαιοσύνη προκειμένου να ε, εκδικαστεί η υπόθεση και θα πρέπει να πούμε ότι η εισαγγελία ε, θεώρησε ότι είναι, αποδεκτή, είναι παραδεκτή αυτή η αγωγή και αφορά υποθέσεις ε, οι οποίες ε, όντως επηρεάζουν τα δικαιώματα και πως αυτός ο αγώνας θα πρέπει να δοθεί. Η αγωγή που καταθέσαμε Αναφορούσε την παραβίαση των δικαιωμάτων και τον καθορισμό των λόγων των ενώσεων που προσέφηκαν στην δικαιοσύνη, την αρμοδιότητα των ε, δικαστικών αρχών. Θα παρακολουθήσω λοιπόν αυτό το πρόγραμμα για να δικαιολογήσω το, το έργο μας. τα πω όλα τα στοιχεία που επελέγησαν, καταχωρήθηκαν ως ε, μυστικά, ως απόρριτα και αφορούν οι δραστηριότητες νέα εταιριών Microsoft 2007, του Yahoo το 2008, Google ε, και Facebook το 2009, YouTube και Skype το 2010, Honeywell το 2011 και Apple το 2012. Το πρόγραμμα Prism επιτρέπει να συλλέξουν στοιχεία αυτών των υπηρεσιών που αφορούν τις δραστηριότητές τους, το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ε, φωτογραφίας, ε, το μεταφορά δεδομένων, καθώς επίσης και της ε, συνομιλίας online. Αυτή η συλλογή δεδομένων γίνεται από και προς το εξωτερικό και αφορά τα εξυπηρετητές η NSA σε μια υποδομή που του επιτρέπει να ε, λαμβάνει όλες τις προφορίες αλλά το γεγονό είναι ότι αν η SA, FBI, DIA, SIA μπορούν να ε, εισέρχονται και να λαμβάνουν ό,τι στοιχεία επιθυμούν τηλεφωνικά, νούμερα τηλεφωνικά, ταυτοποιητές, και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν με, μισό, με 500, με 500 εκατομμύρια συγγνώμη, ε, κοινωνιών προσωπικών που έχουν συλλάξει μέχρι το 2013 είχαν συλλέξει συνολικά 97 δισεκατομμύρια πληροφορίες το Μάρτιο του 2013. Στέιβ Ντόλινγκ, πρόσωπος της ε, Apple, δήλωσε ότι δεν ε, έδωσε ποτέ ε, δυνατότητα πρόσβασης. Αλλά οι Αμερικανικές αρχές λένε ότι το πρόγραμμα Prison ήταν ήδη γνωστό το 2016. 2006, Και ο πρόεδρος Μπάμα δήλωσε ότι αυτό που έχουμε είναι δύο προγράμματα που εξοδοτήθηκαν από το Κογκρέσο και επιβεβαιώθηκαν, επικυρώθηκαν από αυτό. Επίσης, βυρογνώμονες κρίνουν ότι οι εμπλεκόμενες ε, εταιρείε δεν μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίε, ήταν, ήταν υποχρεωμένοι να διαθέτουν ε, τις απαραίτητες δομές. Επίσης δημοσιεύτηκε μια ανακοινωθέν το οποίο λέει ότι δεν μπορούμε να στοχεύσουμε κάποιους αλλοδαπούς αν δεν υπάρχουν ε, ε ουσιαστικοί λόγοι. Αποτέλεσμα ήταν ότι τα στοιχεία τα οποία ε, δημοσιεύθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, παρακαλώ, μήπως μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά. Ναι, slowly, slowly. Προκύπτουν λοιπόν στοιχεία τα οποία έχει δημοσιεύσει ο τύπο, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δημιούργησαν ένα σύστημα συλλογή ιδιωτικών δεδομένων που αφορά τόσο του Αμερικανού πολίτε όσο και ε, τι ε, αλλοδαπέ οργανώσει και ενώσει αυτά τα σύστημα. Λοιπόν, μέσω ε, διαφόρων ε, κλείδων μπορούσαν να ελέγχονται. Και αυτό μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι με, την με το προκάλημα της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος η κυβέρνηση ε, δημιουργεί κάποιους κανόνες ετεροδικίας για να δημιουργήσει ένα σύστημα πάνω, υπεράνω όλων. Σε αυτές τις ε, συνθήκες ε, η οργάνωση τη δική μας θεώρησε ότι ήταν σκόπιμο να ε, προσφύγουν στον εισαγγελέα του Παρισιού προκειμένου μια αρχική έρευνα να ξεκινήσει προκειμένου να χαρακτηρίσει τα παραβιάσεις. Δεύτερον, σχετικά με την ε, θέμα της παραδοχής ε, των ε, αγωγών. Το, άρθρο 2, παράγραφος 2, ο αστικός κώδικας, ο κώδικας αναφέρει ότι η, ότι μία παράβαση αφορά άμεσα τους πληγέντες από μία τέτοια πράξη σύμφωνα με τα άρθρα 6 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης των Δικαιωμάτων και τα 385 του ε, ποινικού κώδικα, το δικαστήριο το 2010, Οκτώβριο 2010 αναφέρει ότι για να είναι παραδεκτή μια τέτοια περίπτωση οι συνθήκες στις οποίες βασίζεται θα πρέπει να επιτρέπουν την ε, άμεση σχέση με μια παραβίαση του ποινικού δικαίου. Το δικαστήριο λοιπόν, όπως έκανε και ο ανακριτής, θεώρησε ότι πολιτική, θα μπορούσε να γίνει δεκτή η πολιτική αγωγή για, την, ε, για θέματα της ε, της παραβίασης ε, κάποιων αρχών, ειδικά σε ό,τι φορά την εκτροπή δημοσίων ε, μέσων, οδηγεί σε μια ε, απειλή των ε, δικαιωμάτων Θεώρησε λοιπόν ότι αυτή η προσφυγή είναι παραδεκτή και έτσι το δικαστήριο υπενθυμίζει ότι οι ενώσεις υπόκεινται στο νομικό, στο ε, δίκαιο της χώρας και τα θέματα που αφορούν οι αγωγές ε, επηρεάζουν πρόκειται για θέματα τα οποία αφορούν την ε, πρόσβαση σε ε, ιδιωτικά δεδομένα, ιδιωτικά στοιχεία. Και η FDA και LDA σου ιδιαίτερα δραστήριες στον τομέα της ιδιωτικότητας και των παραβιάσεων στον ε, τομέα του διαδικτύου κρίνουν ότι αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν την βάση των δράσεων τους. Επίσης, Μήπως μπορείτε να κλείσετε παρακαλώ για να τεθούν και οι ερωτήσεις. Θέλει να κάνει κάποιες συμπερασματικές δηλώσεις. Ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για παραβάσεις τις οποίες έχω ταξινομήσει, θα σας αναφέρω τους τίτλους για να μην μακρηγορήσω. Πέντε παραβάσεις είναι εξίσου. Πρόσβαση και παράνομη διατήρηση, σε ένα, σε ένα σύστημα επεξεργασία δεδομένων η συλλογή ε, και εξαπάτηση ε, τρίτον η απόπειρα ε, παραβίασης ε, ιδιωτικών δεδομένων ε, χρήση και διατήρηση καταγραφών και δοκιμών και, και εγγράφων και τέλος η απόπειρα παραβίασης ε, του δικαιώματος των ηλεκτρονικές ε, συνομιλίες. Είναι γεγονός ότι μπορούμε να βρούμε σε άλλα κάτι, ότι κάτι τέτοιο δεν ε, επιτρέπει να προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, αλλά στην Γαλλία επιτρέπεται και αν τελικά. Ε, σας ευχαριστούμε. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας για να αντιληφθούμε λίγο την ουσία της υπόθεσης. Κύριο Άλμπρεχτ, πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για αυτή την συνολική εικόνα της διαδικασίας που μας δώσατε καθώς επίσης και την άποψή σας σε σχέση με την άσκηση ενδικών μέσων ατομικά. Θα ήθελα να γνωρίζω εσείς τι θα περιμένατε από τα μέλη των κοινοβουλίων στα κράτη-μέλη, καθώς επίσης και από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και από τις κυβερνήσεις όσον αφορά την ατομική αποζημίωση εκείνων που άσκησαν ένδικα μέσα. Ο Πρόεδρος και να προσθέσω και κάτι. συνάδελφοι θα μιλήσουν για την υπόθεση του άρθρου 8 και των ατομικών προσφυγών. Θα ήθελα λοιπόν πριν να, από αυτούς να πω το εξή, να ρωτήσω μάλλον. Ποια υποστήριξη έχει στην διάθεσή του ο τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών. Δηλαδή, σας υποστηρίζει ο κόσμος, έχει την υποστήριξη των μέσων μαζικής ενημέρωση. Πρώτα απ' όλα, για αυτό που με ρωτήσετε, τι περιμένουμε από τους, τους βουλευτές. Περιμένουμε να βελτιωθεί η νομοθεσία και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή να δημιουργηθούν διαδικασίες ελέγχου και διαδικασίες που να περιορίζουν αυτές τις δραστηριότητες. Φυσικά δεν θα κάνουν το ίδιο όλες, όλα τα κράτη, αλλά ε, δεν είναι δυνατόν μία δραστηριότητα να θεωρείται αποδεκτή σε ένα κράτο και όχι αλλού. Αναμένουμε λοιπόν από τους βουλευτές, τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου να κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιωθεί το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά επίσης και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Ε, επίσης να προχωρήσει η προσχώρηση, ε, μάλλον η υιοθέτηση της οδηγίας με βάση την οποία θα γίνεται ο έλεγχος βάσει βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και επίσης περιμένουμε να δοθεί το δικαίωμα της ατομικής προσφυγής, κάτι που ακόμα δεν υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε και από την γαλλική κυβέρνηση. Στη Γαλλία υποβάλαμε αυτήν την προσφυγή. Και δεύτερον, με βάση την απόφαση που θα λάβει η εισαγγελία, η δικαιοσύνη, να εξεταστεί το θέμα συνολικά στη Γαλλία και ε, αργότερα και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίως στις χώρες DCP θα πρέπει να κατά την άποψή μου βελτιωθεί η διαδικασία. Το προαιρετικό πρωτόκολλο στην ΕΣΔΑ θα δώσει το δικαίωμα ατομικής προσφυγής. Θα μπορούσαμε να ε, επεκτείνουμε αυτό το δικαίωμα και στις ε, χώρες ΔΣΕΠΕ. Τώρα όσον αφορά την υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων, εγώ θα μιλήσω εξ τη της ε, Ένωσης Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ΕΛΔΕΑ και η ΕΦΤΕΑ υπέβαλαν από κοινού προσφυγή στηριζόμενη στο εθνικό δίκαιο και στο διεθνές δίκαιο. Θεωρούμε ότι Έχουμε την υποστήριξη του συνόλου των μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά τα, δικαιώματα, τα ψηφιακά δικαιώματα, την προστασία της ιδιωτικότητας στο ίντερνετ στην Γαλλία. Δεν έχει ακόμα όμως λάβει το θέμα τη δημοσιότητα που θα έπρεπε έτσι ώστε να διεξαχθεί μια δημόσια συζήτηση και αυτό ίσως θα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να περιμένουμε και να ζητήσουμε από τη γαλλική κυβέρνηση μια δημόσια συζήτηση. Έχω μια ερώτηση που ίσως είναι τοποθέτηση. Στην έναρξη της τοποθέτησής σας αναφερθήκατε στη Λαμπετούζα και νομίζω αν σας ερμηνεύω σωστά αυτό που θέλατε να πείτε είναι ότι όλες αυτές οι τεχνικές δυνατότητες, όλες αυτές τα συστήματα ελέγχου τελικά καταλήγουν να θεωρούν κάθε πολίτη δυνητικά ύποπτο και ότι όλοι υφίστανται και υπόκεινται σε παρακολούθηση. Και είπατε αν κατάλαβε καλά ότι όλα αυτά γίνονται εξαιτία της τρομοκρατίας. το λοιπόν, μιας και μιλήσατε με τόση σαφήνεια, γίνεται, είναι δυνατόν να είμαστε σίγουροι ότι οποιαδήποτε αναζήτηση ή α, κάποιο profiling που γίνεται με βάση λέξεις κλειδιά θα μπορούσε να είναι σωστή, λέμε ότι ψάχνουμε βελόνα στα άχυρα. Η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Γνωρίζουμε καν τι είδου βελόνα ψάχνουμε. Μήπως όλη αυτή η πλημμυρίδα των μέτρων παρακολούθησης στην πραγματικότητα μας παραπλανούν από το πραγματικό θέμα, το πραγματικό ζήτημα, μήπως εν τέλει δεν είναι ορθά. Αυτό θα είναι το τελευταίο ερώτημα που θα λάβουμε. Ακούσουμε. Αυτό που θα προσθέσω εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα το θέσω και στους άλλους ομιλητές. Από γνωρίζω, στη Γαλλία ε, έχει δοθεί λιγότερη δημοσιότητα στο πρόγραμμα PRISM από ότι στη Γερμανία. Συμφωνείτε? Επίσης η Γαλλική Βουλή πώς αντέδρασε και πώς σχολιάζεται την αντίδρασή της Επίσης, αν μπορούσατε κάπως να μας κατατοπίσετε για τη χρονική αλληλουχία, πώς θα προχωρήσει η διαδικασία από εδώ και πέρα. Τώρα για κυρία Ζήπελ. Ναι, πιστεύω ότι προσανατολίζεται προς την ασφάλεια. Δηλαδή υπάρχουν ε, άτομα τα οποία είναι πιο ε, ε, ελέγχονται περισσότερο από ότι οι άλλοι και σε ό,τι φορά το έλεγχο στα σύνορα είναι το πιο καταστροφική ιδέα μπορούμε να έχουμε σχετικά με το ζήτημα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαθέτουμε μια σειρά τεχνικών μέσων ε, για να κάνουμε αυτό το οποίο αφορά την ε, προστασία του ίντερνετ ε, και όταν πρόκειται για τους φτωχοδιάβολους που προσπαθούν να διασχίσουν τη θάλασσα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Εν ε, δεν υπάρχει κάποιο πρότυπο για διευθέτηση, ρύθμιση αυτών των δεδομένων, ε, αυτών των υποθέσεων και όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενώ έχουμε όλα τα τεχνικά μέσα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αν ε, όλα τα σύνορα ε, παρακολουθούνται, ο κόσμος λέγεται ότι είναι πολύ πιο ασφαλής από ό,τι στο παρελθόν. Εγώ το αμφισβητώ κάτι τέτοιο. Ο έλεγχος με τον οποίο γίνεται, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι και με τον οποίο ε, ακολουθούνται κάποιες ε, ε διαδικασίες πραγματικά αποτελούν προσβολή της δημοκρατίας τώρα την πολιτική της Ελλάδα της ε, Γαλλίας ε, οι αρμόδιοι δουλεύουν και ο τρόπος με, με τον οποίο έχει αντιμετωπίζει το ζήτημα με την μη σύσταση κάποιων εξεταστικών επιτροπών. Πραγματικά η επιτροπή μου, η ομάδα μου, η ένωσή μου, όπως θέλετε πείτε έχει κάποιες ε, αμφιβολίες ε, και όντως ε, κάποιες χώρες άλλες έχουν δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία προς τα ζητήματα αυτά, συμπεριλαμβάνουμε των κύριο πολιτών αλλά και των βουλευτών, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα στη χώρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης ε, για την εδώ παρουσία σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και παρακαλώ παραμείνετε μέχρι το τέλος της ε, συζήτησης. Επόμενος αγορητής ε, είναι ο Νίκ Πίκλος, διευθυντής του Big Brother Watch, οργάνωση που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και στα πλαίσια της προστασίας των μελιωδών δικαιωμάτων και ε, για την ε, ανάπτυξη της Παγκόσμια οικονομίας που θα βασίζεται στο διαδίκτυο τα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι ο στόχος τη Big Brother Watch και ο λόγος της προσφυγής μας δεν είναι να βάλουμε τέλος στην παρακολούθηση, αλλά να διασφαλίσουμε ότι σε ένα δημοκρατικό ε, κράτος η παρακολούθηση είναι προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή με ένα σκεπτικό το οποίο να μπορούν οι πολίτες να ακολουθήσουν και να κατανοήσουν και να εμπιστευτούν. Αυτή τη στιγμή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Οι πολίτε δεν εμπιστεύονται το ε, νομικό πλαίσιο. Τι έκανε ο Edward Snowden. Μα έδειξε δύο πράγματα. Καταρχά την κλίμακα και την φύση τη παρακολούθηση, η οποία είναι ε, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι προβλέπουν οι εθνικέ νομοθεσίε και ό,τι σκόπευαν ε, να ορίσουν οι νομοθέτες. Και δεύτερον, ότι όπου έχουν εκχωρηθεί οι αρμοδιότητες παρακολούθησης, αυτές οι αρμοδιότητες έχουν ε, πέσει αντικείμενο εκμετάλλευση και κατάχρησης και έχουν ε, δημιουργηθεί υπερμεγέθη σε μηχανισμοί παρακολούθησης που έχουν ξεφύγει πολύ από τα όρια ε, που προβλέπει ο νόμος. Τώρα όσον αφορά τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα παραθέματα. Καταρχάς σε κάτι που είπε ο Νάιτζελ Έξτερ, ο πρώην διευθυντής της ε, MI6, είπε ότι αισθάνομαι ότι αυτοί που θα ενδιαφερθούν περισσότερο για τις ε, δραστηριότητες της ε, NSA και των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών δεν έμαθαν και κάτι που δεν ήξεραν. Ο Έντουαρντ Σνόντεν έχει κάνει ένα μεγάλο καλό για, τον, για το κοινό και πιστεύω και ελπίζω ότι θα είναι μόνο η αρχή. Η αρχή μας έδειξε την κλίμακα της παρακολούθησης και την κλίμακα της αδυναμίας των νομοθετών να ελέγξουν τις ε, ε, ενέργειες παρακολούθησης. Ο νόμος εφαρμόζεται με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον ε, οποίο είχε αρχικά συνταχθεί. Ο στόχος είναι η αύξηση της διαφάνειας, κάτι το οποίο είναι κοινό συμφέρον. Είναι πραγματικά ντροπή το ότι μια τέτοια συζήτηση δεν διεξάγεται στην ε, Βρετανία και θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις σας ε, γι' αυτό το θέμα. Ωστόσο, θα ήθελα να σημειώσω ότι παρά την ε, έλλειψη ενδιαφέροντος, όταν άρχισε η νομική διαδικασία. Μέσα σε λίγες μέρες είχαμε συλλέξει υπογραφές από πάρα πολλούς πολίτες και είχαν ενημερωθεί πάρα πολύ από τις, για τις δραστηριότητές μας. Ο κόσμος λοιπόν συζητά για αυτά που κάνουμε. Τα μέσα ενημέρωσης συζητούν και αναφέρονται σε αυτό που κάνουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίσουμε πλέον και δεν μπορεί να γνωρίσει το κοινό. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου έχει εξετάσει τις ε, ε, δραστηριότητες παρακολούθησης, όχι όμως το πρόγραμμα Τέμπορα, το οποίο είναι και το κύριο υπεύθυνο για τις ε, παραβιάσεις ε, που έχουν διαπιστωθεί. Η Επιτροπή Ελέγχου δεν ανέφερε καν το πρόγραμμα Τέμπορα στην έκθεσή της. Και αναρωτιέ, αναρωτιόμαστε εάν δεν ήξερε για την ύπαρξή του ή εάν απέκρυψε τις δραστηριότητές του. Σύμφωνα με το άρθρο 8 πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα στην εφαρμογή των ε, ενεργειών παρακολούθησης ε, και αυτό δεν συνέβη στην περίπτωση αυτή. Αρχικά αυτό που θέλαμε είναι να προσφύγουμε ενώπιον των Βρετανικών δικαστηρίων, αλλά όπως ε, ακούσατε και πιο πριν σχετικά με τα ένδικα μέσα, ε, ναι μεν θα ήταν ε, κάτι που θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς, ωστόσο κάθε προσπάθειά μας να προσφύγουμε σε Βρετανικό Δικαστήριο απερίφθη και βρεθήκαμε ενώπιον ε, απορρίτου. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει κρίνει στην υπόθεση και έναντι ότι τέτοιου τύπου εκδίκαση των υποθέσεων δεν αποτελεί αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί έφεση ε- ε- εναντίον μια υπόθεση που έχει ε, κρυθεί σε, κυκλισμένο το Η τεχνολογία λοιπόν έχει, έχει προχωρήσει με τέτοιον τρόπο που επιτρέπει την αδιάκρηκτη μαζική συλλογή δεδομένων με τρόπο ο οποίος από τη φύση του δεν μπορεί να υποκειται στις ε, νομοθετικές, ε, στο νομοθετικό έλεγχο, δεν μπορεί να είναι αναλογικός, ούτε ε, να συλλέγονται αυτά τα δεδομένα με συγκεκριμένο σκοπό. Έτσι λοιπόν αυτές οι δραστηριότητες θεωρούμε ότι παραβιάζουν το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Καθώς επίσης και την παράγραφο 2 που αφορά στην υποχρέωση των κρατών να σέβονται την ΕΣΤΑ στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Τώρα, ε, έρχομαι στην υπόθεση Brown. Θα σας ζητήσω να διαβάσετε την μαρτυρική κατάθεση, κυρίως το υπόμνημα, στο οποίο λέγεται ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει δημιουργηθεί το σύστημα τεμπόρα είναι, τέμπορα ε, είναι η παρακολούθηση, ο λόγος μάλλον για τον οποίο έχει δημιουργηθεί το σύστημα τέμπορα είναι η παρακολούθηση όλων των δεδομένων τα οποία περνούν μέσα από τις βρετανικές ε, επικοινωνίες. Αυτό που ήδη αναφέρθηκε από ομιλητές είχε σχέση με το ιδιαίτερο στοιχείο του, του βρετανικού νομικού συστήματος. Και αυτό νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει στους πολίτες να καταλαβαίνουν και να είναι αρκετά ξεκάθαρο με ποιον τρόπο υποφασίζονται αυτές οι ε, δραστηριότητες παρακολούθησης, ποιες είναι ασφαλιστικές δικλείδες, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, ποιες κυβερνητικές ε, υπηρεσίες και ποιες ασφαλιστικές δικλείδες μπορούν να τους προστατεύσουν από κατάχρηση αυτών των δεδομένων, καθώς επίσης και έλεγχοι οι οποίοι θα ε, ασκούνται σε αυτές τις κυβερνητικές υπηρεσίες για να διαπιστωθεί ότι δεν παραβιάζουν τις εξουσιοδότηση που τους δόθηκε. Διαφορετικά θα συνεχίσει να αυξάνεται αυτή η μυστική και μαζική παρακολούθηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε την Κωνσταντζε Κότς, η οποία είναι πλήρω, επιστήμων πληροφορικής και εργάζεται στο Ερευνητικό Κέντρο Πολιτισμού και Πληροφορικής. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε και την δική της οπτική γωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα παρουσιάσω μερικά στοιχεία που ενδιαφέρουν αυτήν την Επιτροπή. Στην Επιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων υπάρχουν αυτή τη στιγμή όλες οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές. Τώρα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ε, δυνατότητα που μου δώσατε να τοποθετηθώ για τις ε, πρακτικές ε, που ε, δημοσιεύθηκαν σχετικά τον, από τις Βρετανικές εμιστικές υπηρεσίες και θα αναφερθώ συγκεκριμένα στην παραβίαση της σύμβασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις Αμερικανικές εμιστικές υπηρεσίες. Τους τελευταίους μήνες έχουμε διαπιστώσει ότι δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει μόνο η δυνατότητα παρακολούθησης της ψηφιακής και διαδικτυακής κίνησης, αλλά η δυνατότητα αυτή χρησιμοποιείται κιόλα. Και όχι από δικτατορικά καθεστώτα, αλλά από, την, ε, από κυβερνήσεις της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι στην παρακολούθηση ε, υπερπόντιων καλωδίων και ε, συνδέσεων οπτικών ινών. Αυτή η περίπτωση είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, προσωπικά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ανήκω σε ε, εκείνους ε, τους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν παραβίαση και υπέστησαν υποκλοπή δεδομένων. Υποκλοπή δεδομένων που έγινε στα πλαίσια αυτής της μαζικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Ο κύριος Πίκλ αναφέρθηκε λοιπόν στο Στρασβούργο στην έλλειψη πρόσβαση σε, στοιχεία και στην άρνηση των μυστικών υπηρεσιών να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές. Και οι μόνες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δημοσιεύθηκε από τον Edward Snowden. Επίσης, ούτε η γερμανική κυβέρνηση ούτε και άλλες κυβερνήσεις έχουν δεχτεί να διερευνήσουν επίσημα το θέμα αυτό. Τώρα, πέρα από το αν ήταν δικαιολογημένη η παρακολούθηση αυτή από τις Βρετανικές Εμιστικές Υπηρεσίες για τους ε, λόγους ε, εθνικής ε, ασφάλειας. Το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα και το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών συμπεριλαμβάνεται στην σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. και οι Βρετανικές εμιστικές υπηρεσίες έχουν σύμφωνα με το Βρετανικό ε, δίκαιο όχι μόνο να ε, διεξάγουν υποκλοπές και συλλογή δεδομένων αλλά και να μην εκατονομάσουν ε, τους στόχους τους, τους στόχους τους να μην ενημερώσουν αργότερα τα πρόσωπα τα οποία ε, αφορούσαν αυτές οι υποκλοπές. Τώρα, σύμφωνα με την Βρετανική νομοθεσία, ε, τώρα έχουν ε, ανακοινωθεί από την ε, κυβέρνηση των Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου η πρόθεση για συζήτηση βελτίωσης ε, της ε, προστασίας των πολιτών. Όμως αυτό αναφέρεται στον, στους ημεδαπούς πολίτες και όχι στους αλλοδαπούς. Οι... Στην περίπτωση αυτή έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το Βρετανικό Δίκαιο, να συνεχίσουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται δεδομένα των, πολιτών, ε, των αλλοδαπών πολιτών. Τώρα, υποκλοπές ε, και συλλογή δεδομένων παρατηρήθηκε σε ε, καλώδια οπτικών ινών, 24, 24 κόμβους οπτικών ινών στην υπηρετική Ευρώπη, ακόμα και ενδοευρωπαϊκές συνδέσεις. Τώρα, παραβίαση για εμά δεν καθιστά μόνο η ανάλυση των δεδομένων, αλλά και η συλλογή αυτή. Δεν μας δόθηκαν κανενός είδους πληροφορίες, ούτε σχετικά με το ποιος ε, συνέλεξε τα δεδομένα αυτά, ούτε και εάν υπήρχε κάποια ε, έγκριση και η γερμανική κυβέρνηση δεν ε, ανέλαβε κανένα, καμία νομική ενέργεια για διερεύνηση του περιστατικού αυτού. Αυτό αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Να σας ε, υπενθυμίσω επίσης και την ε, περίπτωση υποκλοπών των, ε, ε, από τις μυστικές ε, υπηρεσίες της Βρετανίας στην Belgacom, τις οποίες πελάτες ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ άλλων. Στην περίπτωση δικτυοπαραβίασης της Belgacom παρατηρήθηκε συλλογή δεδομένων μέσω ενός προγράμματος εξαιρετικά αναπτυγμένου προγράμματος σε δίκτυο παραβίασης. Και εδώ πέρα υπάρχει ξεκάθαρη ε, παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας κάποιου κράτους μέλους του Βελγίου, το οποίο, η κυβέρνηση του οποίου είναι μερικός ιδιοκτήτης της Belgacom. Το πρόγραμμα αυτό συν, ε, είχε να κάνει με την συλλογή δεδομένων κωδικών πρόσβασης και αποκρυπτογράφησης κωδικοποιημένων επικοινωνιών. Όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πελάτες της Belgacom, όχι όμως μόνο εκείνοι. Το ΝΑΤΟ και το SWIFT είναι επίσης ε, οργανισμοί που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Belgacom. Επίσης, να αναφέρουμε και το πρόγραμμα Edge Hill των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, το οποίο είναι παρόμοιο με το πρόγραμμα Bullion της NSA. Με το πρόγραμμα Edge Hill, οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες υποκλέπτουν συστηματικά κωδικοποιημένες επικοινωνίες και τα προγράμματα αυτά δεν έχουν σταματήσει ακόμα και μετά την ε, δημοσιοποίησή τους, ακόμα και μετά την ενημέρωση του κοινού για τις ε, δραστηριότητες αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές ε, είδαμε πώς ενεργούν οι μυστικές υπηρεσίες. Είτε χρησιμοποιούν διάφορα νομικά παραθυράκια, είτε χρησιμοποιούν πληροφοριοδότες οι οποίοι εργάζονται στις, ε, στους παρόχους ε, αυτούς και συλλέγονται και υποκλέπτονται δεδομένα από πολλούς ε, παρόχους, από το Facebook, από το Skype, από την Google και το Yahoo. Αυτή τη στιγμή οι μυστικές υπηρεσίες δεν έχουν κανέναν απολύτως έλεγχο και δρούνε σε μία γκρίζα νομική ζώνη. Γι' αυτό και εμείς προσφύγαμε και πιστεύουμε πέραν αυτού ότι δεν είναι μόνο νομική ευθύνη, είναι και πολιτική ευθύνη να υπάρξει αντίδραση και να υπάρξει κάποιος ε, περιορισμός. Αυτό μπορεί να γίνει για παράδειγμα με ένα σύμφωνο ε, μη επίθεση στο διαδίκτυο καθώς και με μέτρα κατά της ε, δίκτυο Επίσης, να αναφέρω ότι και ο πρώην αρχηγός ε, της NSA ε, και ο νυν ε, επικεφαλής της NSA είπε ότι δεν ψάχνουμε βελόνα στα άχυρα, συλλέγουμε και μαζεύουμε όλα τα άχυρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντζε. Τώρα θα έχει την ευκαιρία να απαντήσει σε ερωτήσεις. Η πρώτη από αυτέ είναι του Άξελ Βό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πίκλη, κύριε Κουρτ για τι παρουσιάσει σα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχά το γιατί ασχολούμαστε περισσότερο με την αμερικανική πλευρά και όχι τόσο με την ε, Βρετανική. Εντάξει, είναι προφανές ότι όταν, αυτά, όταν έγιναν αυτές οι αποκαλύψεις από τον ε, Edward Snowden αφορούσαν κυρίως ε, τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ θα ήθελα εν πάση περιπτώσει να ρωτήσω, εσείς πού βλέπετε τα όρια ή πού θα θέτατε τα όρια ανάμεσα στην ιδιωτική σφαίρα και την δημόσια ασφάλεια στο διαδίκτυο. Έχω την εντύπωση ότι το διαδίκτυο δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιωτική σφαίρα λόγω της ε, ιδιαιτερότητάς του, ότι είναι ένας κοινός ε, δημόσιος χώρος. Εσείς λοιπόν πού θα φετατε όρια, πού σταματα η ιδιωτικότητα και πού αρχίζει η ο δημόσιος χώρος. Επίσης, εσείς που θεωρείτε, από ποιο σημείο και έπειτα θεωρείτε ότι ε, υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων στην απλή συλλογή δεδομένων ή και στην, επεξ, ή στην επεξεργασία του. Παρακαλώ. Η ε, κυρία Κούρτς, όσον αφορά την πρώτη ερώτησή σας για την γενικότερη ασφάλεια στο διαδίκτυο, πιστεύω πως καταρχάς πρέπει να ε, δούμε τα κενά που υπάρχουν στην ε, ασφάλεια, τα ε, διαρθρωτικά κενά, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την καθημερινή μας επικοινωνία. Καταρχάς ε, έχουμε παρατηρήσει ότι οι, Αμερικανικές και Βρετανικές αμυστικές υπηρεσίες ανέπτυξαν λογισμικό το οποίο αποκωδικοποιούσε κωδικοποιημένα δεδομένα ενέργειες αυτές έγιναν εκμεταλλευόμενες σε διάφορα παραθυρά και διάφορα κενά στην ε, ασφάλεια ή ε, όπως είπα πληροφοριοδότες που εργάζονταν στις ε, εταιρείες όπως η οπως ειπα πληροφοριοδοτες που εργαζονταν στις εταιρειες οπως η ακόμη για παράδειγμα. Υπήρξε λοιπόν παραβίαση της δομής των, του διαδικτύου. Επίσης, όπως γνωρίζετε, πάρα πολλά συστήματα ε, πλοήγησης, ε, πάρα πολύ ε, πάροχοι, πάρα πολύ, πάρα λογισμικό, έχουν προβλήματα σχετικά με την ασφάλεια. Και ακριβώς αυτά τα προβλήματα εκμεταλλεύτηκαν οι μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχει αγορά για ακριβώς αυτά τα κενά στην ασφάλεια και οι μυστικές υπηρεσίες έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτή την αγορά. Θα μπορούσε να πει κανείς μάλιστα πως έχουν πληρώσει για να υπάρχουν αυτά τα κενά στην ασφάλεια. Και πιστεύω πως αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί ποινικό αδίκημα. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτησή σας για τα ψηφιακά δεδομένα και πού σταματά η ιδιωτική σφαίρα και πού αρχίζει ο κοινός δημόσιος χώρος. Υπάρχουν κάποια Υπάρχει πιστεύω κάποιος σαφή διαχωρισμός ε, και ο προηγούμενος ε, ομιλητής πιστεύω πως αναφέρθηκε σε αυτό. Αναφέρθηκε στην συλλογή και αποθήκευση δεδομένων για προληπτικούς λόγους, κάτι το οποίο δεν θα, ε, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται πλέον. Γιάννη, έχεις και εσύ μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ πολύ και για τις απαντήσεις σας. Εγώ έχω μία ερώτηση σχετικά με αυτά τα προγράμματα παρακολούθησης. Το Tempora, το Prism και τα παρόμοια ε, προγράμματα, όποιο όνομα και αν έχουν, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές, στοχεύουν σε διαφορετικά δεδομένα. Εγώ όμως, ε, όπως και πολλοί άλλοι, αναρωτιέμαι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ε, με τι μπορούμε να παρομοιάσουμε αυτήν, ε, την, ε, αυτές τις ενέργειες έτσι, στον αναλογικό κόσμο. Είναι κάτι που δεν έχει απαντηθεί πιστεύω και θα ήθελα λοιπόν να ε, μου πείτε επίσης και πώς αυτό επηρεάζει τον πολίτη, πώς αυτό επηρεάζει το άτομο πώς, ε, πώς ε, παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, του πολίτη και της δημοκρατίας με αυτές τις ε, ενέργειες. Η ερώτηση αυτή απευθύνθηκε και στους δύο σας. Πιστεύω πως ε, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, η κλίμακα θα ήθελα να πω ότι η παρακολούθηση δεν είναι κάτι καινούριο. Και τώρα κύριε Βός ε, αναφερθήκατε στην ιδιωτική σφαίρα και στην ε, και στον δημόσιο χώρο. Όμως να σας πω ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα, ε, μια σειρά στοιχείων που παρακολουθούν στοχευμένα μυστικές υπηρεσίες. Όχι, συλλέγουν τα πάντα. Δεν κάνουν προφίλ και σύμφωνα με αυτά τα προφίλ συλλέγουν δεδομένα. Τώρα, το τι αποτελεί εθνικό συμφέρον. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Μάρκ Ζούκερπεργκ είπε ότι μία δυνατή οικονομία αποτελεί εθνικό συμφέρον. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση έχει πελάτες σε όλο τον κόσμο, τότε Τα εθνικά συμφέροντα υπονομεύονται όταν δίνεται προτεραιότητα σε πολίτες ε, ενός συγκεκριμένου κράτους. Τώρα κύριε Άλμπρεχτ, οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων, την επεξεργασία όγκου δεδομένων, να σας πω το εξής. Ε, στην ε, Μεγάλη Βρετανία έχουμε τον νόμο για την ε, ρύθμιση διερευνητικών αρμοδιοτήτων. Και όταν δημιουργήθηκε ο νόμος αυτός, είχαμε... δεν είχαμε οπτικές σύνες, δεν είχαμε τόσο προηγμένη τεχνολογία. Η τεχνολογία που υπήρχε τότε επέτρεπε την συλλογή δεδομένων σε πολύ μικρότερη κλίμακα από ό,τι τώρα. θα ήθελα να κάνω κι εγώ ένα σύντομο σχόλιο για την τελευταία ερώτηση. Ω ε, τεχνικός πληροφορικής, πιστεύω πως οι δυνατότητε που έχουμε σήμερα είναι ε, τεράστιες για ψηφιακή παρακολούθηση και πιστεύω ότι αυτή η μορφή της ε, ψηφιοποίηση των καθημερινών δραστηριοτήτων μα. δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα το αναλογικό. Έχουμε όλοι τώρα τα smartphone, χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο στα πάντα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν τον όγκο των δεδομένων που ε, κινείται τώρα με την αναλογική εποχή και οι ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται ολόνα και μικρότερες και η χρήση του διαδικτύου γίνεται ολόνα και μεγαλύτερη. και οι εξελίξεις που θα έχουμε σε τρία έως πέντε χρόνια θα είναι πολύ μεγάλες. Πρέπει λοιπόν να συζητηθεί το ζήτημα αυτό, διότι η νομική ασάφεια στον ε, χώρο του διαδικτύου θα οδηγήσει σε ανεξέλεκτη παρακολούθησε και ανεκτέλεκτες εξελίξεις. Και να σας πω επίσης ότι οι τελευταίες 53 τρομοκρατικές επιθέσεις που έλεγαν χώρο στις ΗΠΑ ε, δεν ήταν κάτι που οι μυστικές υπηρεσίες δεν κατόρθωσαν να αποτρέψουν όσο και αν ε, παρακολουθούσαν και συλληνέλεγαν δεδομένα. Ναι, η Άννα Γκόμες. Γνωρίζοντας τις επιπτώσεις που, έχει, που έχουν αυτές οι πρακτικές για το μέλλον, εσείς τι θα προτείνατε να ζητήσουμε από τις αρχές μας από όσους χρησιμοποιούν αυτές τις πρακτικές. Αναφέρατε το σύμφωνο μη επίθεση στο διαδίκτυο. Όμως, ποια είναι η αξία του. Τι θα προσφέρει παραπάνω από τους ε, υφιστάμενους νόμους προστασίας δεδομένων ή από την ε, προστασία που παρέχει το διεθνές δίκαιο. θα προσφέρει δυνατότητα περισσότερου κοινοβουλευτικού ελέγχου, ελέγχου του τι συμβαίνει. Θα προσφέρει κάποιο νέο ε, ένδικο μέσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Τι παραπάνω, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία του. Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ, λέει ο τον Νίκ. Ε, το εξής, ε, αν στο, στο Ηνωμένο Βασίλειο και να πω ότι η παρουσίασή σα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και έτσι κι αλλιώς ε, υπάρχει στο διαδίκτυο, οπότε δεν χρειάζεται να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι τη δική σα άποψη, τη δική σα γνώμη για το τι μπορεί να αλλάξει μετά από αυτήν την ε, προσφυγή, μετά από αυτή τη σειρά προσφυγών σε πολιτικό επίπεδο. Στην ε, πρώτη συζήτηση συζητήσαμε τις ενέργειες ε, στην Γαλλία, στη Γερμανία. Εσείς όμως, τι θεωρείτε πως μπορεί να αλλάξει. Αναφερθήκατε στην, ε, ε, στα όρια ανάμεσα στην εθνική ασφάλεια και στην ατομική ελευθερία. Και για το αν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η γραμμή, αυτό το όριο. Πιστεύω όμως ε, πως, ε, για να είμαι ειλικρινής, έχει χαθεί λίγο η μάχη. Εσείς τι προσπαθείτε να επιτύχετε. Διότι για να έχει κάτι πραγματικό όφελος πρέπει να ξεφύγει από αυτά τα περιορισμένα εθνικά όρια μιας έρευνας. Ποιο θα είναι το πολιτικό επίτευγμα εάν δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο από αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι το ανέφερε και η Κόνσταντ. Το θεμελιώδες πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν έχουμε πληροφόρηση, δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Μπορούμε τουλάχιστον να πούμε ότι είναι προ τιμή των ΗΠΑ που αποχαρακτήρισαν κάποια έγγραφα και μπορέσαμε να μάθουμε τι συνέβη. Κάτι το οποίο ανάγκασε τι εταιρείε να ενημερώσουν του πελάτε του για τι δραστηριότητε παρακολούθηση που ε, διεξήγαν. Τώρα. Ακόμα και η Επιτροπή του Κοινοβουλίου εδώ αμφιβάλλει κατά πόσον το νομικό πλαίσιο είναι επαρκές. Αυτό θεωρώ μας δείχνει ότι οι ασφαλιστικέ δικλείδες δεν είναι επαρκεί. Η δυνατότητα ατομικών προσφυγών από τους πολίτε τίθεται με την επιτάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο για πολλούς λόγους. Νομίζω εδώ υπάρχουν δύο σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι περήφανο για το ρόλο και το νομοθετικό του πλαίσιο, για το ρόλο του Κοινοβουλίου και το νομοθετικό του πλαίσιο. Το είχε αναφέρει και ο Υπουργό Εξωτερικών μα, ανέφερε το, τη σημασία που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βρετανία και η κοινωνία των πολιτών. Όμω, νομίζω ότι όλο και περισσότερο υπονομεύεται ο ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό, δεν μα πιστεύουν πια και δεν έχουμε πλέον το ηθικό ανάστημα να ισχυριστούμε ότι αυτό ισχύει. Δεύτερο σημαντικό θέμα είναι ότι πιστεύω ότι ο κόσμος δεν έχει ακόμα καταλάβει ποια είναι η κλίμακα του προβλήματος. Και νομίζω ότι οι προσφυγές στη δικαιοσύνη μπορούν να μας βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό, να μάθει ο κόσμος στη Βρετανία τι συμβαίνει, να μάθει ότι ε, η παρακολούθηση από τις ΗΠΑ είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Και ευελπιστούμε και άλλες χώρες να βγουν στο προσκήνιο και να δημοσιοποιηθεί τι συμβαίνει σε αυτές. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Φαίνεται ότι θα καταφέρουμε να κλείσουμε την ώρα μας. Για όποιος μας βλέπει από το ίντερνετ να πω ότι απλώς εξεπλάγει, γι' αυτό το είπα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννα Άλμπερχ την Πριζή Ζίπολ και κύριο Βος που ήταν παρόντες σε όλες τις δημόσιες ακροάσεις που διοργανώσαμε για το θέμα. Συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ. Μακάρι όλοι οι συνάδελφοι να κάνουν το ίδιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικές τους ομιλίες. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τη Γραμματεία για αυτή την διοργάνωση και της 8ης Δημόσιας Ακρόασης και όλο το προσωπικό επίσης. Κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για να διοργανηθούν αυτές οι ακροάσεις. Δεν είναι κάτι εύκολο. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Νομίζω τελευταία φορά προεδρεύω σε αυτή την επιτροπή, άρα δεν θα έχω άλλη ευκαιρία να σας ευχαριστήσω.